Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση στην έναρξη της συνεδρίασης. Δύο είναι οι λόγοι τη καθυστέρησης. Ο πρώτος ήταν να περιμέναμε περισσότερους συναδέλφους. Αλλά περιμένουμε και τον καλεσμένο μας. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να ξεκινήσουμε. Σας καλωσορίζω θερμά στη συνεδρίαση και σας καλώ να περάσουμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης καλωσορίζοντας ε, και τους ε, καλεσμένους του κυρίου Ντεκάστρο από την Ιταλία. Καλωσορίζουμε τους ε, επισκέπτες που είναι φιλοξενούμενοι ολόκληρης της Επιτροπής Γεωργίας πια και όχι μόνο του κυρίου Ντεκάστρο. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και ελπίζω να αποκομίσετε θετικές εντυπώσεις από τις εργασίες της Επιτροπής. Περνάμε, όπως σας είπα, στο σημείο 4. Συντελεστής αναπροσαρμογής για τις άμεσες ενισχύσεις που προβλέπεται στο κανονισμό 1306 του 2013 για το ημερολογιακό έτος 2015. Δεν είναι κλασική η ε, έκθεση. Την αναλαμβάνει με συμφωνία των συντονιστών ο πρόεδρος, ο υποφαινόμενος και θα ήθελα να σας δώσω μερικές εξηγήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στι 27 Μαρτίου μία απόφαση για την δημοσιονομική πειθαρχία ε, με βάση τον κανονισμό που προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει κάθε χρόνο να προτείνει στα πλαίσια της εφαρμογής του Μηχανισμού Δημοσιονομικής Πειθαρχίας την σύσταση αποθεματικού κρίσης για τη γεωργία. Αυτό κάνει λοιπόν κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στα πλαίσια της συναπόφασης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν χρόνο προθεσμία μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2015 προκειμένου για να προτείνουν και να ορίσουν το συντελεστή δημοσιονομικής πειθαρχίας. Αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θέσει από μόνη της αυτό το συντελεστή με ε, εκτελεστικό κανονισμό. Στην τελευταία συνεδρία, οι συντονιστές ε, αποφάσισαν να, ε, να εφαρμόσουν την διαδικασία του άρθρου 50 και μου ανέθεσαν ως πρόεδρο την έκθεση αυτή, την γραμματότηση αυτή που είναι εξαιρετικά σύντομη και μάλιστα ε, υποβάλλεται χωρίς τροπολογίες. Αυτή την έκθεση σας υποβάλλω τώρα και με βάση τη διαδικασία θα πρέπει να προβλεφθεί παρόλα αυτά μια προθεσμία για τις τροπολογίες. Αυτή είναι μέχρι τις 7 Μαΐου, 12 το μεσημέρι. Αλλά θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στο εξή, κάτι που είναι και ασυνήθιστο και το συμφωνήσαμε με τους συντονιστές. Ε, ε, καλό θα ήταν ε, και εσείς τα συναυτοί να μην καταθέσετε τροπολογίες, ώστε να μπορέσουμε ήδη να καταλήξουμε σε συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Άλλωστε και το Συμβούλιο δεν πρόκειται να καταθέσει καμία τροπολογία. Αυτό δεν επηρεάζει την ουσία του πράγματος, γιατί ούτως ή άλλως είναι αυτόματος ο υπολογισμός αυτού του συντελεστή αναπροσαρμογής. Απλώς έτσι το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαφυλάσσουν τα προνόμια τους ε, ως ε, μέλο της συναπόφασης, αντί να αφήνουν αυτό το, αυτή την εξουσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επαναλαμβάνω, μέχρι τις 7 Μαΐου υπάρχει προθεσμία για τις τροπολογίες, 12 το μεσημέρι και ελπίζουμε, όπως φάνηκε και στους ε, συντονιστές, ότι δεν θα κατατεθούν τροπολογίες. Η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα γίνει στην πρώτη Ολομέλεια του Ιουνίου. Αν δεν έχετε παρατηρήσεις και σχόλια, δεν ξέρω αν ο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής θέλει το λόγο. Φαντάζομαι όχι. Ο κύριο Ροπέ. Ευχαριστώ, κύριε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράττω με τις ευκαιρίες μια που συζητούμε το θέμα των άμεσων πληρωμών για να σας ευστήσω την προσοχή στην ε, διαφορά που ουσιαστικά παρατηρείται στις διάφορες χώρες από τις άμεσες πληρωμές. Οπότε, μια που το συζητούμε το θέμα αυτό, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι η διαφορά των άμεσων πληρωμών που, έχουν, ε, που είναι, είναι μεγάλη ανά κράτος μέλος. Οι βαλτικές χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Λιθουανίας, την οποία εγώ εκπροσωπώ, ε, είμαστε, ε, παίρνουμε το μικρότερο ποσοστό σε άμεσες πληρωμές και πρέπει να έχουμε υπόψη ότι οι δικοί μας οι γεωργοί έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ από το ρωσικό εμπάργκο, κυρίως στον τομέα του γάλακτος. Θα θέλαμε βεβαίως να σας ε, ευχαριστήσουμε για τη στήριξη από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, αλλά αυτά ουσιαστικά τα χρήματα κάλυψαν τις απώλειες των πρώτων τεσσάρων μενών του 2014. Το εμπάργκο όμως συνεχίζεται και οι απώλειες αυξάνονται. Η παραγωγή γάλακτος δεν κερδίζουν πια τίποτα από την παραγωγή τους και πρέπει να προετοιμαστούν και για τη νέα ε, για τη νέα ε, ε, σεζόν και μπορεί κάποιοι να τα παρατήσουν γιατί δεν τους συμφέρει πλέον. Είχαμε και τον αυθόδη πυρετό, επηρεάστηκαν χώρους όπως η Πολωνία, επηρεάστηκαν, επηρεάστηκε ο τομέας των πουλερικών. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία που έχουμε και θα ενθάρρυνα την Κομισιόν να υποστηρίξει τους γαλακτοπαραγωγούς των βαλτικών χωρών. Τους ή άλλως έχει υπάρξει τέτοια ε, υπόσχεση εκ μέρους του. Ευχαριστώ. Κυρία Σένορα. Ναι. Μια διαδικαστική ερώτηση. Εγώ είμαι καινούρια στην Επιτροπή και στο Κοινοβουλίο. Και μερικές φορές ε, αργό να συλλάβω γιατί πράγμα μιλάμε. Τις προάλλες, όταν στους συντονιστές συζητήσαμε για αυτό το σχέδιο χωρίς τροπολογίες, εγώ είχα ήδη πολλές εμφιβολίες και θέλω τώρα να ρωτήσω τη γραμματεία από νομική σκοπιά αν εμείς οι συντονιστές μπορούμε να λάβουμε μια απόφαση να μην τροποποιήσουμε ένα κείμενο όταν ε, από νομική σκοπιά οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής έχει δικαίωμα να υποβάλει τροπολογίες. Μπορείτε να μου ξεκαθαρίσετε νομικά τι ισχύει. Ε, Πρώτα να δώσω το λόγο και στον ε, συνάδελφο της Γραμματείας. Ήταν σύσταση, δεν ήταν απόφαση αυτή. Η κυρία Σράερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ να μην καταθέσουμε τροπολογία. Αλλά θα πρέπει αυτό να το καταλάβουν ε, όλοι και ιδιαίτερα οι γεωργοί. Γιατί όπως είπε και η προλαλήσασα, ε, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι παίρνουμε τη σωστή απόφαση. Γιατί έχουμε και το ρωσικό εμπάργκο. Θα πρέπει να ξέρουμε τι μπορούμε και τι δεν επιτρέπεται να κάνουμε στην Ευρώπη. Και θέλω να ξέρω όλες τις δυνατότητες που έχουμε για τα θέματα αυτά, για να ξέρω τι μπορώ να κάνω και ποιο είναι το καθήκον μου ως Ευρωβουλευτής, για να μπορώ να το εξηγήσω και στους ε, συμπολίτες μου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα απαντήσω στην ερώτηση της κυρίας Σενσένρα που είναι νομιμή. Πρέπει να είναι σαφές ότι το δικαίωμα κατάθεση τροπολογίας ανήκει σε κάθε βουλευτή και εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή. Γι' αυτό ακριβώς ο Πρόεδρος είπε ότι έχουμε προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών μέχρι τις 7 Μαΐου. Υπάρχει λοιπόν τέτοια προθεσμία και φυσικά κάθε βουλευτή έχει το αναφέρετο δικαίωμα να καταθέσει τροπολογίε. Απλώ ε, ε, το άρθρο αυτό του βασικού κανονισμού έχει ω εξή. Ε, αν κατατεθούν τροπολογίε και θετηθούν και πάμε μέχρι την Ολομέλεια, τότε θα είμαστε σε μια κατάσταση που δεν θα μπορούμε να συμφωνήσουμε σε πρώτη ανάγνωση με το Συμβούλιο που περιμένει ότι δεν θα υπάρχουν τροπολογίε προ υιοθέτηση μέχρι τι 30 Ιουνίου. Έτσι λοιπόν το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Απλώς αυτό το ποσοστό θα έχει υιοθετηθεί από την Κομισιόν με εκτελεστική πράξη. Μπορεί να θεωρηθεί κάτι παράξενο, εδώ είναι και η Κομισιόν, ίσως θα μας το επιβεβαιώσει, αλλά ακριβώς αυτό προβλέπει ο βασικός κανονισμός. Δηλαδή, αν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν καταλήξουν σε συμφωνία μέχρι τις 30 Ιουνίου και μόνος τρόπος να καταλήξουν συμφωνία είναι χωρίς να υπάρχει καμία τροπολογία, η Κομισιόν ε, με εκτελεστική πράξη θα προβεί υιοθέτηση. Στο Συμβούλιο θεωρείται με σαφήνεια ότι θα ε, πρέπει την ε, αρμοδιότητα να την έχει ο συνομοθέτης, γι' αυτό μας πρότειναν αυτή την προσέγγιση. Τώρα, αυτό είπαν και συντονιστές, αλλά και πάλι, για να απαντήσω, κυρία Σέρα, ναι, το δικαίωμα κατάθεση τροπολογιών είναι να το δικαίωμα του κάθε βουλευτή. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ενημερωθήκαμε και μπορούμε να διαμορφώσουμε εμπεριστατωμένα άποψη. Πέραμε τώρα στο σημείο 5 που προβλέπει ανταλλαγή απόψε με τον κύριο Φερνάντες που είναι ο Γενικός Συγητής για τον προϋπολογισμό του 2016 στα πλαίσια της ε, δημοσιονομικής διαδικασίας για το επόμενο έτος. Κατά την έναρξη της ε, δημοσιονομικής διαδικασίας ο Γενικός εισηγητή για τον προϋπολογισμό του 2016 επισκέπτεται τις ε, επιτροπές, τις κοινοβουλευτικέ επιτροπές ε, για ανταλλαγή απόψεων ε, σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητε του προϋπολογισμού για τον επόμενο χρόνο. Φέτος ορίστηκε γενικό εισηγητή ο κύριος Φερνάντε. Τον καλωσορίζω θερμά στη συνεδρίαση τη Επιτροπής και ε, θα ήθελα να το δώσω το λόγο για να μας παρουσιάσει τη δημοσιονομική διαδικασία, τα βασικά χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού για το 2016. Η Επιτροπή θα υποβάλει το, το σχέδιο προβλέψεων ε, μέχρι τα τέλη του Μαΐου για τον προϋπολογισμό του 2016 και θα ήθελα να συνδέσουμε το σημείο 5 με το σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Ο Ζαν Πολ Ντενανό είναι ο συντάκτης της γνωμοδότης Επιτροπής Γεωργίας για το σημείο 6 που προβλέπει τον προϋπολογισμό του 2016. Πρώτα θα δώσω το λόγο στον καλεσμένο μας, τον κύριο Φερνάντες. Και μετά στον συντάκτη της γνωμοδότησής μας, τον κύριο Ντενανό. Παρακαλώ κύριε Γενική Συγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω για τις προτεραιότητες που υιοθετήθηκαν ήδη στην Ολομέλεια, τις κατευθυντήριες ε, γραμμές, τις γραμμές προσανατολισμού, αλλά κυρίως για να ακούσω και τις συμβουλές σας, οι κατευθυντήριες γραμμές. Εκεί έχουμε κάποιες πολιτικές προτεραιότητες που είναι πολύ απλές, αλλά νομίζω και σημαντικές. Μιλάμε για τα τρία ε, στα γαλλικά απασχόληση, επιχείρηση και επιχειρηματικότητα. Και για το στόχο αυτό, φυσικά υπάρχουν σημαντικά προγράμματα όπως ορίζοντες 2020, το COSME, το Erasmus πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων αλλά επίσης έχουμε και ως προτεραιότητα την εσωτερική αλληλεγγύη. Και επί της εσωτερικής αλληλεγγύης η συνοχή αλλά και η γεωργία είναι σημαντικές, η αλία. Δεν ξεχνάμε και την εξωτερική αλληλεγγύη. Και αυτό έχει να κάνει με τον τομέα 4. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τι συμβαίνει γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την αναπτυξιακή βοήθεια, την ανθρωπιστική βοήθεια. Και όλα αυτά σχετίζονται με το στόχο μας ε, που είναι η ασφάλεια. Μιλάμε για τις πληρωμές, ε, τα θέματα πληρωμών ε, θα επιληθούν φέτος ή τουλάχιστον θα προσδιορίσουμε την πορεία που θα ακολουθήσουμε. Έχουμε ακόμα επιχειρησιακά προγράμματα που δεν έχουν τέθει σε εφαρμογή. Ελπίζουμε ότι φέτος όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα θα είναι σε εκτέλεση σε όλες τις χώρες. Κάνουμε λόγο για τον προπολογισμό του 2016. Πρέπει λοιπόν να σεβαστούμε τις δεσμεύσεις μας και πρέπει να σεβαστούμε και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο που έχουμε θετήσει για το χρονοδιάγραμμα. Το σχέδιο προπολογισμού της Κομισιόν θα παρουσιαστεί στις 27 Μαΐου. Έχουμε και το σημαντικό θέμα των προπερασκευαστικών δράσεων και των πιλωτικών προγραμμάτων. Η Κομισιόν, συγγνώμη, η Επιτροπή Γεωργίας αυτή τη στιγμή δεν έχει πιλωτικά προγράμματα σε εκτέλεση. Η προθεσμία είναι 4 Ιουνίου για να παρουσιαστούν αυτά τα πιλωτικά προγράμματα ή οι δράσεις. 4 Ιουνίου επαναλαμβάνω και 17 Ιουνίου είναι η προθεσμία για ε, την υιοθέτηση των εκθέσεων για το τριμερή διάλογο 22-23 Ιουνίου κατόπιν και στην Ολομέλεια θα πάμε τον Ιούλιο στις 3 Σεπτεμβρίου κατάθεση προθεσμίας ε, τροπολογιών δημοσιονομικού χαρακτήρα ε, για τις επιτροπές 17 Σεπτεμβρίου για τις πολιτικές ομάδες ε, και 28-29-30 Οκτωβρίου ψηφοφορία για τις τροπολογίες 12 και 13 Οκτωβρίου ψηφοφορία για το ψήφισμα και κατόπιν ψηφίσουμε στην Ολομέλεια και στα τέλη Οκτωβρίου έχουμε την συζήτηση για τον εισηγητή. Η Γεωργία έχει σημαντικό βάρος στον προϋπολογισμό. Το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και εντός της νέας φιλοσοφίας θα πρέπει να το δούμε ως ένα ταμείο που είναι συμπληρωματικό των άλλων ταμείων της πολιτικής συνοχής και μάλιστα και το θέμα της εφιούς ανάπτυξης θα πρέπει να το αντιληφθούμε εντό αυτού του ταμείου. Φυσικά η βιώσιμη ανάπτυξη είναι κάτι που συμπεριλαμβάνει τα πάντα. Πρέπει να δούμε και το θέμα του ρωσικού εμπάργου. Όμως ε, για Φέτος κάναμε τροποποιήσεις ε, για το γάλα, ε, για τα φρούτα δεν ε, εγκρίθηκαν οι τροποποίησεις αυτές, όμως φυσικά αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ ευαίσθητα για μένα και πρέπει να δούμε και τι συμβαίνει στον τομέα του γάλακτος, γιατί υπάρχει ένα σοβαρός αντίκτυπος λόγω του συστήματος ποσοστώσεων σε ό,τι αφορά την απασχόληση, την προτεραιότητα για την απασχόληση. Και η γεωργία φυσικά πρέπει να είναι εντός. Έχουμε το στόχο της απασχόλησης των νέων. Και αυτός ο στόχος είναι σημαντικός και εντός της γεωργίας. Επιμένω στο θέμα των πιλωτικών προγραμμάτων που θα μπορούσαν να είναι σημαντικά και στην ημερομηνία της 4ης Ιουνίου καθώς αποτελεί την προθεσμία για την παρουσίαση αυτών των πιλωτικών προγραμμάτων. Σε ό,τι αφορά τώρα ε, το χρηματοδοτικό πλαίσιο για το ε, ΦΕΑΓ, για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων. Ε, ουσιαστικά προβλέπεται κάτι ανώτερο σε σχέση με αυτό που θετήθηκε στον προπολογισμό του 2015, αλλά φυσικά πρέπει να ακούσουμε την πρόταση για το σχέδιο προπολογισμού της Κομισιόν που θα παρουσιαστεί στις 27 Μαΐου και για το Γεωργικό Ταμείο, για το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ε, στον προγραμματισμό Έχουμε μια μικρή μείωση, δεν είναι πολύ σημαντική, αλλά όπως σας είπα, περιμένουμε στις 27 Μαΐου να δούμε το σχέδιο του προϋπολογισμού που θα μας παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να ακούσω και τις δικές σας συμβουλές και περιμένω φυσικά και σχόλια από τον εισηγητή σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Φερνάντες. Ο κύριος Δενανό τώρα για να μας παρουσιάσει τη δική του άποψη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με προσοχή το Γενικό Εισηγητή, ο οποίος επισήμανε κάποια προβλήματα και αν το Κοινοβούλιο κάθε χρόνο αποφαίνεται επί της δημοσιονομικής χρήσης, παρόλα αυτά έχει περιορισμένο περιθώριο λιγμών, γιατί έχουμε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, παρόλο που ίσως έχουμε και μια διάμεση αναθεώρηση και πρέπει φυσικά να τηρούνται οι κανόνες της δημοσιονομικής πειθαρχία. Ε, στην γνωμοδότησή μου δυστυχώς δεν έχω συγκεκριμένα ποσά, γιατί ακόμη δεν έχουμε λάβει το σχέδιο προϋπολογισμού. Αν δεν κάνω λάθος, στις 27 Μαΐου θα υποβληθεί, οπότε λίγος χρόνος αναμονής μας έχει μείνει. Και η Επιτροπή Προϋπολογισμών, θα, στην οποία είμαι και μέλος, ε, όπως και ο κ. Φερνάντες, θα εξετάσει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το σχέδιο προϋπολογισμού. Παρόλο που δεν έχουμε συγκεκριμένα ποσά, συγκεκριμένους αριθμούς, από τη μέχρι τώρα ε, πείρα μου, θα ήθελα να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Τρεις είναι οι γενικές παρατηρήσεις. Πρώτη, αφορά το γενικό προπολογισμό της κοινή γεωρικής πολιτικής. Η ΚΑΠ είναι από τις σημαντικότερες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα η πιο ολοκληρωμένη από τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Εξασφαλίζει την ασφάλεια των τροφίμων μας, την επιστηστική μας ασφάλεια, συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και τίνει προς μία αηφορία, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει, όπως είπε ο κύριος Φερνάντε, ε, την αύξηση της απασχόλησης σε πολλές περιοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα πρόσφατα είχαμε μεταρρύθμιση της ΚΑΠ για να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι συμβάλλουν στη χρηματοδότηση της κοινή γεωρικής πολιτικής. Και στην γνωμοδότησή μου ζητώ η χρηματοδότηση της ΚΑΠ να μείνει τουλάχιστον στο τωρινό της επίπεδο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αποθεματικό της κρίσης, το ποσοστό αυτό συντελεστή ε, που περιλαμβάνεται στον κανονισμό για τη δημοσιονομική προθε... πειθαρχία είναι 1,39 και κάτι τεκατό. Είναι το σύνηθε ποσοστό. Ε, βέβαια αυτό σημαίνει ότι θα μειωθούν αντίστοιχα οι άμεσες ενισχύσεις. Αν δεν ενεργοποιηθεί το 2016 αυτό το αποθεματικό κρίσης, ε, ζητώ εννοείται τα ποσά που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί να επανέλθουν στο κονδύλιο των άμεσων ενισχύσεων. Επίσης, ό,τι αφορά τα περιθώρια στη στήλη 2, στη δημοσιονομική χρήση του 2016 θα πρέπει να έχουμε κάποια περιθώρια ε, και να χρηματοδοτηθούν από την υπερισφορά για το γάλα. Ε, γιατί ε, κάποιες χώρες έχουν πρόσφατα ξεπεράσει τα ποσοστό, τις ποσοστώσεις τους γαλακτοκομικές εν ώψη της κατάργησης των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων. Ζητώ λοιπόν αυτά τα έσοδα να παραμείνουν στην γεωργία γιατί είναι μεγάλες οι ανάγκες της και οι γεωργικές μας αγορές υφίστανται ακόμη τις ε, συνέπειες του ρωσικού εμπάργου που δεν πρόκειται να έρθει ο ονούπο, πλήττει πολλούς τομείς. Έχουμε και το ζήτημα του γάλακτος, η αγορά γάλακτος εξακολουθεί να είναι εύθραυστη και ιδιαίτερα μετά τις εξέλιξεις ποσοστώσεις δεν αποκλείεται και μια επιδείνωση της αγοράς γάλακτος. Και συχνά έχουμε και υγειονομικές κρίσεις με σοβαρές πολλές φορές συνέπειες. Η τελευταία ήταν ε, το παράσιτο ξυλέλα φαστιδιώσα στη Νότιο Ιταλία που έπληξε τα ελαιόδεντρα. Κάτι που θέτει σε κίνδυνο τη γεωργία μας. Ένα σημαντικό ζήτημα που έθεσε ο κύριος Φερνάντες είναι η ανάπτυξη της υπαίθρου, η αγροτική ανάπτυξη σημαντικός πυλώνας της ΚΑΠ. Και ως πρώην, πρόεδρος, ως περιφερειάρχης παρακολούθησε την εφαρμογή του Λίντερ πολύ σημαντικό και στο πρόγραμμα για την Ήπεθρο και την διαφύλαξη θέσεων εργασίας στην Ήπεθρο. Αυτός ο δεύτερος πυλώνας της ΠΑΚ, η αγροτική ανάπτυξη, είναι συμπληρωματικός και όπως είπε ο κύριος Φερνάνδης συμβάλλει στην εδαφική συνοχή. Πολύ σημαντικό θέμα. Επίσης, ε, ιδιαίτερη σημασία προσδίδουμε στην ε, εγκατάσταση στις γεωργικές δραστηριότητες νέων γεωργών. Γιατί αν δεν έχουμε μια ανανέωση γενναιών θα εξαφανιστούν ε, οι γεωργοί στην Ευρώπη και θα χαθεί η γεωργία μας. Γι' αυτό και είμαι υπέρ των ενασμάτων στους νέους γεωργούς προκειμένου να εξασφαλίσουμε αηφόρο γεωργία και μάλιστα με οικονομικές, οικολογικές ε, και κοινωνικές επιδόσεις. Γι' αυτό και θα ήθελα να προβλεφθούν επαρκή κονδύλια για να αντισταθμιστεί το πρόβλημα της αστάθειας των αγορών, που είναι πρόβλημα που μαστίζει όχι μόνο την αγορά γάλακτος, αλλά και αγορές άλλων προϊόντων. Επίσης, ε, οι πιλωτικές δράσεις είναι πολύ σημαντικές. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τη διαφάνειά τους και να βελτιώσουμε τη θέση των παραγωγών στην ε, επιστηστική αλυσίδα. Γιατί ένα προϊόν ε, έχει χαμηλό κόστος παραγωγής και χαμηλή τιμή παραγωγής, αλλά στα ράφια των σούπερ μάρκετ η τιμή του τριπλασιάζεται, τετραπλασιάζεται για να μην πω ακόμη χειρότερα. Επίσης, έχουμε ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, τα απορροκυπευτικά και το γάλα στα σχολεία. Το υπερψηφίσαμε πρόσφατα στην Επιτροπή Γεωργίας. Προτείνω μία μικρή δημοσιονομική αύξηση, 20 εκατομμύρια για το πρόγραμμα αυτό, προκειμένου να ευθυγραμμιστούμε με την ψηφοφορία στην Επιτροπή Γεωργίας. Αυτό το συμπλήρωμα θα επιτρέψει τα κράτη-μέλη που εφάρμοσαν σωστά αυτό το πρόγραμμα να συνεχίσουν ε, να απολαμβάνουν ένα σημαντικό κονδύλιο και να συνεχίσουν να το εφαρμόζουν. Γι' αυτό θέλω μία μικρή ενίσχυση του προγράμματος. Επίσης, θα ήθελα να στηρίξουμε ιδιαίτερως τη μελισσοκομεία. Πολύ σημαντικός κλάδος η μελισσοκομεία, γιατί όχι μόνο εξασφαλίζει την αυτάρκειά μας ε, και την επάρκειά μας σε μέλη, αλλά συμβάλλει στην ε, βιοπικιλότητα με την κατάλληλη γονιμοποίηση, επικονίαση. Είναι σημαντικό λοιπόν να στηρίξουμε και τη μελισσοκομεία. Ευχαριστώ και σημείωσα και την ημερομηνία της 14ης Ιουνίου που είπατε κύριε Φερνάντες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να τονίσω κάτι που είπατε κι εσείς στην αρχή της ε, παρουσίασής της, ότι το αποθεματικό της κρίσης που δεν έχει χρησιμοποιηθεί με βάση τον συντελεστή αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων, όσα κονδύλια δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από το αποθεματικό κρίσης, να επιστρέψουν στον κορβανά των άμεσων ενισχύσεων για την επόμενη χρονιά και να μην χρησιμοποιηθούν για άλλους στόχους. Γιατί πρώτα χρησιμοποιούνται άλλα κονδύλια και το αποθεματικό θα είναι ή το ίστατο μέτρο. Αλλά σε καμία περίπτωση θα πρέπει λόγω του αποθεματικού να μειωθούν οι άμεσες ενισχύσεις. Πολύ σωστά το είπατε και το επισημάνατε και εγώ υπερθεματίζω. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Σλάιερ. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήταν και η χτεσινή ε, συζήτηση που κάναμε πολύ ενδιαφέρουσα ε, και ευχαριστούμε Πρόεδρε για το περιεχόμενο που δώσατε. Τώρα παρακολουθούμε τη δεύτερη, ε, το δεύτερο κομμάτι αυτής της συζήτησης και το θέμα των κονδυλίων. Βεβαίως το μέσο του γάλακτος είναι στην πρώτη θέση, Βεβαίω έχουμε και τον, το θέμα των πουλερικών, του χειρίου κρέατος, των φρούτων. Είναι πολλοί οι τομείς που έχουν επηρεαστεί και βεβαίω οι γεωργοί παντού στην Ευρώπη ε, πλήττονται. Ε, συμφωνώ λοιπόν ε, για το θέμα αυτό. Χτες μιλήσαμε για το τι είναι, ποια είναι τα χρήματα που θα μπορούσαν τελικά να υπάρξουν για τους Γιώργους. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει ένα μεγάλο βάρος όμως προς τους γεωργούς. Τους μιλάμε συνέχεια για την ευζοία των ζώων, υπάρχει οδηγία για το νερό, υπάρχει ο ένας κανονισμός που καταλήγει τελικά να τους αφορά και το ερώτημα είναι μπορούμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τέτοια πιλωτικά προγράμματα δεν λέω ότι πρέπει να τα καταργήσουμε, αλλά είναι σωστό να, να προσφέρουμε αυτά τα προγράμματα στους ε, γεωργούς. Τελικά τους βοηθούμε, γιατί οι πολυεθνικές είναι αυτές που αναλαμβάνουν τελικά όλες αυτές τις ε, δραστηριότητε. και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εγώ το λέω κάθε μέρα. Ε, πολλοί γεωργοί πραγματικά ε, ουσιαστικά κόβονται δευτερά τους από όλα αυτά τα διοικητικά εμπόδια που τους βάζουμε μέσω της νομοθεσίας που ψηφίζουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή και για τις πρώτες του προτάσεις. Ουσιαστικά μπορούμε να τις στηρίξουμε, τις ε, χαιρετίζουμε. Και σε σχέση με την χθεσινή ακρόαση μπορώ να πω ότι ε, αυτή ε, η μαγική λέξη που λέμε πάντα, η μείωση της γραφειοκρατίας πρέπει να συνεχίσει να μας εμπνέει. Ε, Βεβαίω πρέπει να συνεχίσουμε τη μεταρρύθμιση γεωργική πολιτική και για τη διαχείριση από την πλευρά κράτου αλλά και για του ίδιου του ε, γεωργού. Έχουμε, έχουν φυσικά ε, δικαίωμα οι Γεωργοί να καταλαβαίνουν την ε, γεωργική πολιτική που τους αφορά και έτσι όπως την προωθούμε νομίζω ότι δεν την καταλαβαίνουν πια γι' αυτό καταλήγουμε σε προβλήματα. Επίσης να πω ότι υποστηρίζω το θέμα αυτό του αποθεματικού για τις κρίσεις. Ε, πρέπει όντως αν δεν χρησιμοποιείται το αποθεματικό όπως γίνεται καμιά φορά να μπορεί να μεταφερθεί στην επόμενη χρονιά. τις ε, κρίσεις συνήθω δεν μπορούμε να τι προβλέψουμε, απλώ γίνονται, συμβαίνουν και όταν υπάρχουν κάπω πρέπει να τις διαχειριστούμε. Οπότε καλό θα ήταν αν μπορούσαμε να έχουμε έτσι ένα αποθηματικό στην άκρη για να μπορέσουμε να τι αντιμετωπίσουμε. Γιατί βεβαίω τα προβλήματα αναφέρονται και στην έκθεση. Ούτως ή άλλως είχαμε και παλαιότερα προβλήματα. Έχουμε και τώρα ένα έξτρα πρόβλημα με, τους, ε, με το ρωσικό εμπάργκο. Για του νέου γεωργούς δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κάτι που ήθελα να πω όμω είναι το θέμα των, ε, του, του, των φρούτων και του γάλακτος στα, ε, στα σχολεία. Είναι μεγάλη ευκαιρία αυτή και οι συνάδελφοι μου είπαν ότι ε, θα υπάρξει μια τέτοια πρωτοβουλία, να υπάρξει ένα πιλωτικό πρόγραμμα παρόμοιο για, τους, για τα σχολεία. Αλλά η Γεωργία πώς μπορεί εδώ πέρα να εμπλακεί. Στα σχολεία μπορεί να εμπλακεί. με το διατροφικό μοντέλο, ας πούμε, που θα προωθηθεί, που θα εφαρμοστεί στα σχολεία. Και βεβαίω ε, μπορούμε έτσι να προωθήσουμε και την περιφερειακή ε, γεωργία. Δεν υπάρχει καλύτερο από αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε λοιπόν αυτό μέσω της, ε, του προγράμματος αυτού για τα φρούτα και, τα, και το γάλα στα σχολεία. Πρέπει λοιπόν αυτό το πρόγραμμα να το προωθήσουμε έτσι ώστε να, να μην έχει τόση πολύ γραφειοκρατία. Εγώ έχω, ε, έχουμε κάποιες επιλογές, έχω συζητήσει πολλές με διαφόρους διευθυντές σχολείων. Μπορούμε να πάμε να, πούμε, να αγοράσουμε το γάλα κατευθείαν από τον γαλακτοπαραγωγό είναι πιο φτηνό προφανώς ε, για μένα. Αλλά αυτό μπορεί να μην μπορεί να μπει στο ε, πρόγραμμα το ευρωπαϊκό. Ε, εκεί λοιπόν είναι το πρόβλημα. Να φύγει η γραφειοκρατία από τη μέση. Συμφωνούμε με το πρόγραμμα είναι καλό, αλλά η εφαρμογή του είναι πραγματικά πάρα πολύ γραφειοκρατική και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία που έχουμε έτσι ώστε από την επόμενη χρονιά να γίνει η, γεωργία, πολιτική για τη γεωργία πιο φιλική προς, τον, προς τους γεωργούς. Προς τον παρόν έχουμε έναν ε, πόλεμο χαρτιού ε, από την νομοθεσία και τα λοιπά που ψηφίζουμε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό για να μην ε, χάσουμε τις ευκαιρίες που έχουμε απλώς και μόνο λόγω γραφειοκρατικών κανόνων. Γιατί στο τέλος δεν θα μπορούμε να προχωρήσουμε τα προγράμματα που θέλουμε. Και είπα ήδη, έχουμε το θέμα των ποσοστώσεων που αυξάνονται. Γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις ως προς αυτό, ε, ως προς τον έλεγχο γιατί πάντα αυτό είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό, αλλά ε, ε επίσης ε, η, τα ποσοστά του λάθους αυξάνονται και αυτό είναι σημαντικό. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε και να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει, νομίζω εγώ τουλάχιστον, γιατί προς το παρόν ακριβώς είναι πάρα πολύ μεγάλη η γραφειοκρατία. Εμείς έχουμε μια πολύ, αγαπάμε πάρα πολύ την, ε, τη γερμανική γραφειοκρατία γιατί θεωρούμε ότι είναι η καλύτερη του κόσμου αλλά στέλνουμε τόσα πολλά χαρτιά και εντολές στους γεωργούς που μας λένε ε, δεν, δεν καταλαβαίνουμε καν τι γράφουν αυτά τα χαρτιά, πώς θέλετε να τα εφαρμόσουμε. Και δύο χρόνια μετά έρχεται ο ελεγκτής και ξέρει ότι κάτι έχει γίνει λάθος και προφανώς ε, εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα. Από αυτή λοιπόν την οπτική το θέμα αυτό θα πρέπει να το λύσουμε. Πρέπει να αποφεύγουμε ε, λάθη. Πρέπει να μειώσουμε τη γραφειοκρατία. Και πρέπει και στο πρόγραμμα για το 2016 αυτό να αποτελέσει τον πυρήνα του, ε, των προσπαθειών μας. Αυτό θα πρέπει να είναι στον πυρήνα. Η, ε, η μείωση της γραφειοκρατίας. Και ελπίζω να το καταλάβουν τελικά και οι γεωργοί ότι όντως μειώνουμε τη γραφειοκρατία. Ευχαριστώ. Χθε είχαμε εκτενή συζήτηση με θέμα την απλούστευση της κοινή πολιτικής και τη μείωση της γραφειοκρατίας και ένα τμήμα της ε, ομιλίας σας αφορούσε τη χθεσινή μας συζήτηση. Ο κύριος Φεράν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ είμαστε οι υπερομανοί πυροσβέστες, δηλαδή από μηχανισμούς από την ε, Κομισιόν, όπως το παθηματικό της κρίσης, για να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις και βλέπουμε ότι δεν επαρκούν, όπως μας είπε και ο εισηγητής, ε, σε ό,τι αφορά το ρωσικό εμπάργκο και οι συνέπειες επίσης είναι ε, βαριές στους περισσότερους αγροτικούς τομείς. Επίσης, το θέμα δεν είναι η αλληλοβοήθεια εδώ, αλλά υπάρχει κακό πολιτικό όραμα, γι' αυτό δεν αρκούν ε, ε, τα αποθεματικά. Έτσι λοιπόν ε, πρέπει να ε, θέσουμε με διαφανή και γρήγορο τρόπο το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα αποθεματικά της ε, κρίσης. Ε, θα πρέπει όταν δεν έχουν δαπανηθεί τα κονδύλια να πάνε στους γεωργούς. Επίσης, τα κονδύλια που αφαιρώνονται στην γεωργία έχουν μειωθεί σχεδόν 20% τα τελευταία 15 χρόνια σε συνεχή και σήμερα δεν θέλουμε να τα δούμε, να μειώνονται ακόμη περισσότερο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σένερα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω κάποιες προτεραιότητες που θα ήθελα να συμπεριληφθούν στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπάρχει υποστήριξη στις ε, μικρές ε, εκμεταλλεύσεις γιατί νομίζω ότι δημιουργούν πολλές θέσεις εργασίας, ε, φροντίζουν το περιβάλλον, είναι πάρα πολύ σημαντικές για να αποφύγουμε μία μάστιγα που είναι οι δασικές πυρκαγιές και ιδίως στη χώρα μου, στην Καλήσια, πραγματικά κάθε χρόνο έχουμε τεράστιες απολύσεις σχόλια. Θα ήθελα επίσης να συμπεριλάβω μεταξύ των προτεραιοτήτων την πρόθεση και τη διάθεση των τοπικών αγορών ε, και ε, των δραστηριοτήτων που συμβάλλουν ε, στην δίσδυση των αγορών αυτών ε, σε τοπικό επίπεδο. Επίσης, συμφωνώ με τόσο είπε ο για τη στήριξη της μελισσοκομείας. Θα ήθελα και εδώ να συμπεριλάβουμε την καταπολέμηση των κάποιων απειλών, όπως παραδείγματο χάρη είναι η χρησιμοποίηση φυτοφαρμάκων κτλ. Η κυρία Ράνς Γκαρσία. Ευχαριστώ. Εγώ με ιδιαίτερη ικανοποίηση αντιμετωπίζω την αφορά που γίνεται στο γαλακτοκομικό τομέα ως υπεύθυνη της πολιτικής μου ομάδας ε, για την μεταρρύθμιση ε, στον τομέα του γάλακτος. Ανισχούμε πάρα πολύ για το τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Έχει υποθεί από την Επιτροπό ότι είναι πολύ θετικό το μέλλον, όμως εμείς βλέπουμε να υπάρχει πολύ μεγάλη αβεβαιότητα για το γαλακτοκομικό τομέα. Έτσι λοιπόν ε, καλώς ορίζουμε οποιαδήποτε βοήθεια μπορεί να δοθεί στον τομέα αυτή τη στιγμή. Επίσης, στήριξη στη μελισσοκομεία είναι σημαντική για ε, την ε, δουλειά που κάνουν ε, οι μέλισσες και φυσικά οποιαδήποτε ενίσχυση για το πρόγραμμα διανομής φρούτων και γάλακτος στα σχολεία είναι ευπρόσδεκτο γιατί οι νέοι και τα παιδιά είναι το μέλλον μας και καθώς είναι και τα παιδιά είναι το μέλλον μας και δεδομένου ότι ο κύριος Γιάρα αναφέρθηκε στις προθέσεις μου για την παρουσίαση ενός πιλωτικού σχεδίου εγώ θα ήθελα να σας πω ότι στα πλαίσια αυτών των προγραμμάτων σχεδόν ποτέ δεν έχουμε αγροτικού χαρακτήρα προγράμματα και εγώ θα προτείνω ένα που είναι απαραίτητο γιατί αν τα παιδιά είναι το μέλλον μας σας παρουσιάζω ένα πρόγραμμα πρόγραμμα έτσι ώστε οι νέοι και τα παιδιά να λάβουν κατάρτιση και ενημέρωση για τα ποιοτικά εργαλεία των ε, γεωργικών προϊόντων, ε, τα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών, ε, είτε το περνούν στα ψηλά, είτε δεν κάνουν καμία αναφορά στις γεωγραφικές ενδείξεις, στην ονομασία προέλευσης, στις παραδοσιακές ποικιλίε και φυσικά πρέπει να τα μάθουν αυτά τα πράγματα τα παιδιά γιατί όταν γνωρίζουν τις ετικέτες, ξέρουν τι σημαίνουν, μπορούν να τις διαβάσουν, τότε βοηθούν στο να μπουν ευκολότερα τα προϊόντα αυτά στα σπίτια τους. Αυτό έγινε, παραδείγματο χάρη, με το κάπνισμα, όταν ε, τα παιδιά άρχισαν να λένε στους γονείς να σταματήσουν να καπνίζουν. Ε, έτσι έχουμε μικρότερο αριθμό καπνιστών σήμερα. Έτσι λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι η γνώση είναι σημαντικό εργαλείο για την υποστήριξη. Εδώ μπορούμε να μιλάμε πάρα πολύ για τις ετικέτες των γεωγραφικών ενδείξεων, για τις ονομοσίες προέλευσης, για τις γεωγραφικές ενδείξεις, όμως μένουμε μεταξύ μας και μόνο εμείς τα γνωρίζουμε. Πρέπει να κάνουμε αυτή την προσπάθεια για να τα διαδώσουμε αυτά και τα παιδιά να διαβιβάζουν αυτές τις πληροφορίες στο σπίτι τους. Στα 28 μέλη, όπως σας είπα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα είτε το αναφέρουν στα ψηλά ή ούτε καν αναφέρουν αυτό το τόσο χρήσιμο εργαλείο για την ευρωπαϊκή οικονομία και για την υγεία των ευρωπαϊκών καταναλωτών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρόντε. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για το θέμα των κρίσεων, νομίζω ότι είναι αρκετά αρνητικό αυτό που έχουμε να κάνουμε. Ε, εγώ είμαι από τη Δανία και στη Δανία υπάρχει μια τάση να καταδικάζουμε πολύ γρήγορα τη γεωργία. Και παρόλο που κάποιοι μιλούν για τη γεωργία, πολλοί ε, κόσμος θα πει γιατί να έχετε εσείς ένα έξτρα ταμείο για την ε, κρίση. Υπάρχουν και άλλοι που πλήττονται από κρίσεις. Επίσης, τα μέτρα για την κρίση είναι ουσιαστικά, προκύπτουν ουσιαστικά από τις ε, άμεσες πληρωμές. Από εκεί θα προέλθουν τα τα κονδύλια. Οπότε ουσιαστικά είναι σαν να κλέβουμε προσπαθώντας να βάλουμε χέρι σε, αυτό το, σε αυτά τα κονδύλια για τις ε, κρίσεις. Και αυτό πρέπει να ε, το εξασφαλίσουμε ότι δεν πρόκειται να γίνει και να είναι σαφές σε όλους. Σε ό,τι αφορά τώρα συγκεκριμένη βοήθεια για μικρούς γεωργούς, κατανοώ απόλυτα την ε, διαρθωτική πρόσβαση σε ό,τι αφορά τα όσα είπαν οι συνάδελφοι. Αλλά πρέπει να πω ότι η γεωργική μας πολιτική θα πρέπει να προωθεί ανταγωνιστική γεωργία. Αν δεν έχουμε ανταγωνιστική γεωργία στην Ευρώπη, ουσιαστικά θα πληρώσουμε ένα πολύ υψηλό τίμημα σε αυτόν τον παγκοσμιοποιημένο κόσμο με το ελεύθερο εμπόριο, το οποίο κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος. Ανταγωνιστική γεωργία λοιπόν, θα αυτή θα πρέπει να είναι η επικεφαλίδα, σε αυτό θα πρέπει να ε, επικεντρωθούμε. Βεβαίως μέσα στις δομές που ήδη υπάρχουν από τις, ε, στις διάφορες χώρες. Και φυσικά με σεβασμό στους ε, μικρούς γεωργούς. Τώρα, σε αφορά τη γραφειοκρατία. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να τα χαλάσουμε όλα. Ε, κάναμε μια ακρόαση χτες. Ε, ας ξεκινήσουμε εμείς από εδώ. Κάθε φορά που υπάρχει μια νομοθεσία από το Κοινοβούλιο, έχουμε τα ψηλά γράμματα, έχουμε πάρα πολλές λεπτομέρειες ε, και καταλήγουμε τελικά με ένα κείμενο το οποίο ουσιαστικά εμποδίζει τον, τον καθένα που το διαβάζει να καταλάβει ποια θα είναι η πρακτική του εφαρμογή και η πρακτική του επίπτωση σε... όταν θα εφαρμοστεί. Και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το να, είμαστε, να το δούμε πολύ προσεκτικά στην Επιτροπή μας, αλλά και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Έχουμε μεγάλη ευθύνη εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο και για τη δική μας τη γεωργική πολιτική και για τους κανόνες των επιδοτήσεων που είναι τόσο αδιαφανείς. Τέλος, σε, σχέση με τα όσα είπε ο κύριος Γιάς για το γάλα στα σχολεία και τα φρούτα. Με όλο το σεβασμό για την Ολρίκη ε, Μούλερ, η οποία είναι εισηγήτρια από τη δική μου την ομάδα. Εγώ είμαι πραγματικά πολύ σκεπτικό για το πρόγραμμα αυτό. Στη δική μου τη χώρα, λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τρελή. Ε, μπορεί όντως να έχουμε καλή πρόθεση με αυτές τις ε, πρωτοβουλίες, αλλά πρέπει να δούμε τελικά πού αποσκοπούν όλα αυτά. ακούμε από τη μία ότι ε, ταΐζουμε ουσιαστικά τα νέα παιδιά και από την άλλη διευρύνουμε τέτοια προϊόντα που περιέχουν, ε, διευρύνουμε τα προγράμματα με τέτοια προϊόντα που έχουν πάρα πολύ υψηλή περιεκτικότητα στη ζάχαρη. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό που θέλουμε τελικά να πετύχουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χάιτεμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Οι προλαλήσαντες έχουν δίκιο. Τα κοινοτικά κονδύλια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς μας στην παγκόσμια αγορά. Τα, κονδύλια αυτά, τα κοινοτικά κονδύλια θα πρέπει να επενδύουν στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία ώστε απότερος σκοπός μας να γίνει να αποκτήσουμε κάποια αυτάρκεια και να μην εξαρτώμαστε συνεχώς από την βρυξελιώτικη γραφειοκρατία. Δεύτερον, για την ίδια την έκθεση. Πιστεύω ότι τον γαλακτοκομικό τομέα τον αναφέραμε παρκώς, γιατί δεν είναι ο μόνος που επλήγει από το ρωσικό εμπάργο και άλλοι τομεί έχουν θυγεί. Και κάποιοι γεωργοί που εκτρέφουν και πουλερικά για παράδειγμα και αυτοί αξίζουν ενίσχυσης. Ο γαλακτοκομικός τομέας ήδη λαμβάνει αρκετές ενισχύσεις με, τη, με το καθεστώς της τρεματικής ενίσχυσης. Να αναφερθούν και άλλοι τομείς, να μην περιοριζόμαστε μόνο στο γαλακτοκομικό. Πριν δώσω το λόγο στον επόμενο μιλητή, θα ήθελα να καλωσορίσω τους επισκέπτες ε, του κυρίου Χόισλινγκ από τη Γερμανία. Καλώς ήρθατε. Ο κύριος Ροπέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που οι εισηγητές ε, επισήμαναν ε, τα κέρια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο γαλακτοκομικός τομέας, ιδιαίτερα από το ρωσικό εμπάργο. Εγώ θα επικεντρωθώ σε άλλα θέματα. Η ενίσχυση έχει στόχο την, την επιβίωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Αν αδρανίσουμε, μερικές ε, γεωργικές επιχειρήσεις θα χρεοκοπήσουν. Θα πρέπει αυτή την ευθύνη να την αντιμετωπίσουν σοβαρά τα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά το αποθεματικό της κρίσης, οι σωστές αποφάσεις ελήφθησαν το 2014 όταν ε, το αποθεματικό της κρίσης ε, συστήθηκε από τις άμεσες ενισχύσεις. Είμαι υπέρ της κοινοτικής θέσης. και της αυστηρότητάς μας απέναντι στη Ρωσία θα μπορούσαμε να είμαστε ακόμη πιο αυστηροί και απαιτητικοί και τα, τα προβλήματα του ρωσικού εμπάργου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με κονδύλια από τις άμεσες ενισχύσεις για να μην αφήσουμε τους γεωργούς στη μοίρα τους. Σε ό,τι φορά το πρόγραμμα για το γάλα. Το 1 τρίτο των σχολείων ε, δεν χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα. Αν όλα τα σχολεία χρησιμοποιούσαν το πρόγραμμα για το γάλα, θα εξανεμίζονταν πολύ γρήγορα τα κονδύλια. Σε ό,τι αφορά τώρα τον αυθόδη πυρετό των χείρων στις βαλτικές χώρες. Τι κονδύλια θα αφιερωθούν και από πού θα προέλθουν για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα στις Βαλτική. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ριμπέιρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέει κυρία Ριμπέιρο, καταρχήν σε σχέση με το σχέδιο που μας ε, παρουσίασε συνάδελφος Εράνς, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για διάφορους λόγους καταρχήν, γιατί σήμερα είναι της μόδας ε, τα fast food ε, και με εύκολη πρόσβαση και είναι και πιο φθηνά. Και έτσι λοιπόν εμείς ε, φυσικά δεν θέλουμε τα παιδιά μας ε, να τρώνε κάτι τέτοια, προϊόντα αλλά θέλουμε να τρώνε γεωργικά προϊόντα και φαίνεται ότι ε, δεν υπάρχει ουσιαστικά κάποια αντίφαση με το πρόγραμμα διανομής φρούτων και γάλακτος στο σχολείο. Επομένως πρέπει να το υποστηρίξει αυτή η Επιτροπή το πρόγραμμα αυτό. Κάτι άλλο για το γαλακτοκομικό τομέα εδώ αναφέρθηκε και ότι ήδη δέχεται ενισχύσει ο γαλακτοκομικό τομέα και ότι ε, δεν ε, μπορούμε να μην αναφέρουμε τις ορεινές περιοχές ε, και τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές. Ποινικοποιήθηκαν πάρα πολύ οι περιοχές αυτές, ιδιαίτερα στο γαλακτοκομικό τομέα. Έχουμε δει μεγάλη μείωση στις τιμές του γάλακτος που πληρώνονται στον παραγωγό. Έτσι λοιπόν πρέπει να δημιουργηθεί ένα ταμείο που να προστατεύει τους γεωργούς μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, μια υπερισφορά ε, η οποία ε, σχετίζεται με τις χώρες που είχαν ποσοστό πέρσι να μπορεί να απορροφηθεί από το Γενικό Προπολογισμό της ε, Κομισιόν ε, και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργηθεί ακριβώς αυτό το τομείο που θα προσφέρει ασφάλεια στους γεωργού, έτσι ώστε να μην ε, βλέπουμε εμείς κάθε φορά να υπάρχει τέτοια μείωση στην τιμή που πληρώνεται στον παραγωγό. Ο κύριε Σεμπάστια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι για τα όσα άκουσα σε σχέση με το πώς κάποιοι από τους ε, μηχανισμούς μας ε, ε, δεν λειτουργήσαν έτσι όπως έπρεπε, όπως οι μηχανισμοί για την αντιμετώπιση του ρωσικού εμπάργου. Ε, θα ήθελα να δώσω έμφαση στον τομέα των ε, οποροκυπευτικών. Είναι ένα θέμα στο οποίο αναφέρεται και η έκθεση του κ. Μελό που θα εγκρίνουμε το απόγευμα η Ευρώπη δεν παράγει επαρκή προκυπευτικά και ε, βλέπουμε ταυτόχρονα ότι εγκαταλείπονται πάρα πολλά εκτάρια και εκμεταλλεύσεις κυρίως στην Νότια Ευρώπη που παρήγαγαν αυτά τα προϊόντα. Αυτό σημαίνει ότι ο δίκτυπος των άμεσων ενισχύσεων και τη στήριξη στην παραγωγή αυτή δεν λειτουργεί. Έτσι λοιπόν βλέπουμε μεγαλύτερη ε, εξάρτηση από το εξωτερικό στον ε, διατροφικό τομέα και βλέπουμε ότι μειώνεται και η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών ε, και μάλιστα αρχίζουν αυτά τα προϊόντα να θεωρούνται πολυτελή και μάλιστα και λόγω της λιτότητας ε, πολλές οικογένειες δεν μπορούν να τα καταναλώσουν. Έτσι λοιπόν ε, δίνουμε έμφαση προκειμένου αυτό το σχέδιο διανομής φρούτων στο σχολείο να εφαρμοστεί ε, από τους δικούς μας θεσμούς με την απαραίτητη όθηση και να διασφαλίσουμε ότι όλα τα κράτη θα δώσουν ενισχύσεις και στον τομέα των φρούτων και λαχανικών. Και δυστυχώς στην Ισπανία, παραδείγματος χάρη, που είναι μία από τις μεγαλύτερες χώρες παραγωγούς, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Και τώρα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Διευθυντή Χόισλερ από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Παρακαλώ κύριε Διευθυντά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σχολιάσω έτσι γενικά την, την πρόταση κειμένου για το πρόγραμμα για το 2016. Προφανώς όλες οι παρεμβάσεις είναι προσωρινές, το είπε και ο εισηγητής. Η επίσημη υποβολή της πρότασης θα γίνει στις 27 Μαΐου. Το 2016 θα είναι το έτος όπου θα εφαρμοστεί πλήρως η μεταρρύθμιση και σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά της στοιχεία. Δηλαδή, για πρώτη φορά θα υπάρχουν όλες οι αποφάσεις οι οποίες θα εφαρμοστούν σε σχέση με την απόφαση αυτή σε ό,τι αφορά τις δαπάνες. Το 2015 έγινε η σύγκληση, αλλά το 2016 θα είναι πραγματικά το ε, έτος σταθμός γιατί θα υπάρξει μεταφορά των διαφόρων στοιχείων μεταξύ των δύο πυλώνων. Και βεβαίως ε, εκεί θα, κατα, ανεφερθεί και το ποσό που θα λάβει κάθε χώρα, θα υπάρξει η ε, κατάργηση της, ε, των ποσοστώσεων κτλ. Για, τις μετα, τη μεταρρυθμίσεις τώρα, για την ελεύθερη συνδεδεμένη ενίσχυση, κάποια κράτη-μέλη θα δούνε το όνομά τους στο αντίστοιχο κομμάτι της πρότασης και βεβαίως υπάρχουν και άλλα σημεία για, την, για τις άμεσες πληρωμές, ας πούμε, για την Κροατία, την Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Επίσης, ε, θα υπάρξει μικρότερη ε, ανάγκη για κονδύλια για το 2016 και λόγω του ότι θα υπάρξουν υψηλές δαπάνες για τη, λόγω της κρίσης της Ρωσίας ε, το 2015, αλλά προς το παρόν δεν θα υπάρξουν επιπλέον, δεν θα χρειαστούν επιπλέον κονδύλια για το 2016. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι η μέση ζήτηση για την χρηματοδοτική διόρθωση θα εφαρμοστεί μόνο για το αποθεματικό για τις κρίσεις, την οποία το οποίο μάλλον συζητήσετε πιο πριν. Και ένα σύντομο ακόμη ε, σχόλιο για, το, για τη χρηματοδοτική πειθαρχία. Προφανώς ε, τα, με, τα κονδύλια τα οποία δεν θα χρησιμοποιηθούν, αν δεν χρησιμοποιηθούν δηλαδή για μια κρίση, θα μεταφερθούν στο επόμενο ε, έτος και θα επιστραφούν στους γεωργούς θα θυμάστε κάποιους, ε, κάποιες χρονιές ε, που δοθήκαν πάρα πολλά χρήματα στους ε, γεωργούς λόγω μη χρήσης των κονδυλίων. Αυτά τα ποσά λοιπόν και πάλι θα επιστραφούν στους γεωργούς. Σε ό,τι αφορά τώρα το Ταμείο για την Ανάπτυξη Πέθρου. Οι ε, αναλήψει υποχρεώσεων εκεί συνάδουν με τι ε, διατάξει για το σε δημοσιονομικό πλαίσιο για το 2016 και όπω αυτό τα ορίζει. Σε ό,τι αφορά τώρα τι υποχρεώσει πληρωμών για την ε, ανάπτυξη πέθρου, εδώ βρισκόμαστε εδώ και λίγο καιρό σε μια αρκετά τεταμένη κατάσταση. Ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολο ε, αυτές τις υποχρεώσεις πληρωμών της ε, Κομισιόν να τις καλύψουμε στο σύνολό τους και το 2016 αυτή η ένταση θα συνεχιστεί. Ξέρετε ότι το 2016 και για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 αλλά και για το τελευταίο κομμάτι των προκαταβολών και των ενδιάμεσων πληρωμών για το 2014-2020 πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Βεβαίω θα λάβετε πολύ περισσότερες λεπτομέρειε ε, για, ε, για το σχέδιο κειμένου στις 27 Μαΐου όταν θα υποβληθεί επισήμω και φυσικά θα είμαστε στην ε, διάθεσή σα για να σα δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειε για κάθε γραμμή του προπολογισμού. Ακούστηκαν κάποια σχόλια μονομένα για να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένος για τα φρούτα και τα γάλα στο σχολεία. Ζήτησαν κάποιοι βουλευτές να διευρυνθεί το κονδύλι αυτό. Για να σας θυμίσω όμως ότι υπάρχει ένα ανώτατο όριο στην βασική πράξη. Ο νομοθέτης δηλαδή έχει ορίσει πόσο είναι το ανώτατο ποσό που μπορεί να δοθεί ε, για αυτό το πρόγραμμα. Οπότε προφανώς το δημοσιονομικό πρόγραμμα μόνο σε, αυτό το, σε αυτή την νομοθετική πράξη μπορεί να βασιστεί και δεν μπορεί να παρεκκλίνει. Άλλη μία σύσταση για τα πιλωτικά προγράμματα και την προετοιμασία των δράσεων ακούστηκε από πολλούς ευρωβουλευτές. Ε, περιμένουμε τις δικές σας προτάσεις ε, φυσικά. Ξέρετε ότι θα, εξεταθεί, θα εξεταστούν από την ε, Κομισιόν οι δυνατότητες να εφαρμοστούν όλα αυτά το 2016. Αυτά πρόεδρε από μένα και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δύο λόγια να πω κι εγώ πριν ξαναδώσω το λόγο στους εισηγητές μας. Η κοινή γεωργική πολιτική έχει πάρα πολλούς στόχους. Καταρχήν, εξασφάλιση γεωργικού εισοδήματος και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, όπως επισήμαναν και οι συνάδελφοι. Και αυτό με επενδύσεις και με έμφαση στην καινοτομία και ιδιαίτερα στο πλαίσιο του TIP και έχει κάποιους σκοπούς περιβαλλοντικούς ταυτόχρονα η γεωργία, η κοινή γεωργική πολιτική. Υπάρχει ένα στοιχείο όμως ε, κοινωνικό και διαπαιδαγωγικό, για παράδειγμα το γάλα στα σχολεία ή τα απορροκυπευτικά, φρούτα και λαχανικά στα σχολεία. Και υπάρχει και το έκτακτο πρόβλημα του γαλακτοκομικού ε, τομέα και τι θα απογίνει η αγορά μετά την κατάργηση των ποσοστώσεων. Ε, που είναι αρκετά περίπλοκο το θέμα. Α, είδα όμως ότι και ο κύριος Νίκολσον ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπατε υπάρχουν ε, πολλές δυσκολίες ε, που αντιμετωπίζουμε στον τομέα της γεωργίας ε, και στις εκμεταλλεύσεις και στη δική μου περιφέρεια ποτέ δεν έχω δει τα πράγματα να είναι τόσο άσχημα. Έχουμε μεγάλη μείωση των τιμών και το γάλα δεν είναι καλό, ούτε το βόλιο όλα πάνε άσχημα και αυτό το λένε και οι Γεωργοί και υποθέτω ότι η αλήθεια είναι ότι η κοινή γεωργική πολιτική, ο προπολογισμό δηλαδή, για την ΚΑΠ ε, συνεχώς μειώνεται σε ποσοστό αν το δούμε σε αναλογία με το συνολικό προϋπολογισμό της Ευρώπης και αυτό συμβαίνει εδώ και πολύ καιρό και από ό,τι φαίνεται δεν ε, πρόκειται να αλλάξει. Εμεί προσπαθούμε να υπερασπίσουμε τον προϋπολογισμό όσο καλύτερα μπορούμε και φυσικά πάντα προσπαθούμε και προσπαθήσαμε και το Σεπτέμβριο όταν ήταν επίτροπος εδώ να προστατεύσουμε τη γεωργία. Εμένα η δική μου θέση είναι να προστατεύσουμε τον εφιστάμενο προπολογισμό, αυτό που έχουμε εντός ε, του σημερινού πλαισίου και φυσικά ε, ακούσαμε ότι διαφορετικά θα αφαιρούσαμε χρήματα από τη Γεωργία για να χρηματοδοτηθούν ε, άλλα project ε, στην Ευρώπη. Εγώ θέλω να πω ότι αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο. Παραδείγματο χάρη, μετά την ε, κρίση του 2009 είχαμε ε, τεράστια κέρδη που προέκυψαν από τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα οποία δεν επανεπαρδίθηκαν στον ε, τομέα της γεωργίας. Δεν πρέπει να κάνουμε και πάλι το ίδιο λάθος όταν ο γαλακτοκομικός τομέας είναι ιδιαίτερα σταθής και θα πρέπει τα πρόστιμα προκύπτουν από την υπερισφορά να μείνουν εντό του κλάδου ή τουλάχιστον εν γέννη στον τομέα τη γεωργία. Αλλά προπολογισμό για τη γεωργία δεν ήταν βέβαιο και πάντα δύναμη αυτή τη Επιτροπή. Εμεί ε, αντιμετωπίσαμε πέρσι ε, την εξή κατάσταση, δηλαδή το αποθεματικό τη ε, κρίση να έχει χρησιμοποιηθεί για ανθρωπιστικού λόγου και έμειναν πάρα πολύ χρήματα να αντιμετωπίσουμε τι επιπτώσει του ρωσικού εμπάργκο και άλλα που μπορεί να προκύψουν πάντως. Οι δαπάνες ε, για τη γεωργία φυσικά ε, πρέπει και να επικρίνονται. Χτες ακούσαμε κάποιους εμπειρογνώμονες για την απλούστευση της κοινή γεωργικής πολιτικής ε, και το κόστος της διοικητικής πολυπλοκότητας. Έχουμε πραγματικά ε, πραγματικές αλλαγές ε, που μπορεί να γίνουν. Ε, Παραδείγματο χάρη, αν μειώσουμε του έλεγχου που γίνονται από τι εθνικέ αρχέ, θα μπορούσαν τα χρήματα να στοχευτούν καλύτερα αλλού και φυσικά η λιτότητα έχει οδηγήσει τους ε, ανθρώπους στην Ευρώπη να ε, αναρωτιούνται αν έχουμε ε, αξία έναντι των χρημάτων που δίνονται στη Γεωργία. Εγώ νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο και οι εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφεραν δισεκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013 και έχουν δοθεί πάρα πολλές ε, ευκαιρίες για θέσεις εργασίας στο γεωργικό τομέα. Έτσι λοιπόν, ας ε, μην κάνουμε περαιτέρω περικοπές, ας ε, βασιστούμε και ας σε αυτά που έχουμε και ας συμφωνήσουμε με τον εισηγητή ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε τον προπολογισμό στη Γεωργία στο σημερινό επίπεδο. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι ακούσαμε ένα φάσμα επιχειρημάτων χρήσιμα όλα αυτά για το έργο των δύο εισηγητών. Θα δώσω τώρα το λόγο στους δύο εισηγητές. Πρώτα στον κύριο Φερνάντες. Ευχαριστώ. Και αυτό που ακούσαμε δεν έρχονται σε αντίφαση με τις δικές μου αρχικές προτάσεις. Γι' αυτό και χαίρομαι για τη σύμπνοια. Φυσικά δεν πρόκειται να λύσουμε το πρόβλημα της γραφειοκρατίας στον προπολογισμό του 2016. Μπορούμε όμως να το επισημάνουμε και να αφήσουμε κάποια μηνύματα ως προς αυτό. Και ενδιαφέρον θα ήταν ε, σε πολλά προγράμματα να γίνουν μελέτες και να δούμε για να φτάσει ένα ευρώ στον δικαιούχο πόσο έχει στοιχήσει η πορεία του. Μπορεί να μας ε, ευνηδιάσει και να μας καταπλήξει το κόστος που θα έχει αυτό το ευρώ. Και πολλές φορές φταίμε και εμείς, γιατί αντί να απλοποιούμε, περιπλέκουμε. Και αυτό συμβαίνει γιατί διαπιστώνουμε ένα μεγάλο κόστος, αλλά μερικές φορές μειώνουμε και την εκτέλεση προγραμμάτων γιατί οι δικαιούχοι αποθαρρύνονται. Βλέπουν ότι είναι τόσε πολλέ οι προϋποθέσεις που θεωρούν ότι δεν αξίζει τον κόπο να υποβάλουν αίτηση. Ουσιαστικά ενθαρρύνονται οι δικαιούχοι να μην χρησιμοποιούν τα προγράμματα. Και αυτό ισχύει για τα φρούτα, τα λαχανικά. Και να πω και το εξή. Θυμάμαι πέρυσι είχαμε 125 εκατομμύρια με δημοσιονομική γραμμή για το ρωσικό εμπάργκο. Μόνο 37 εκατομμύρια χρησιμοποιήθηκαν από αυτά. Υπάρχει πρόβλημα εκτέλεσης λοιπόν του προϋπολογισμού. Θα πρέπει να δούμε και τους λόγους ε, της μη εκτέλεσης. Γιατί μερικές φορές οι λόγοι της μη εκτέλεσης οφείλονται στην ε, δυσκολία πρόσβασης ε, των δικαιούχων στο πρόγραμμα. Σε ό,τι αφορά το αποθεματικό της κρίσης, δεν ξέρω αν το θέμα αυτό θα αναφερθεί στην διορθωτική επιστολή που περιμένουμε για τα τέλη του έτους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την έγκριση του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου δεν συμφωνήσαμε το αποθεματικό κρίσης ε, να αφαιρεθεί από τα κονδύλια της Γεωργίας. Και δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να το χρησιμοποιήσουμε το αποθεματικό της κρίσης. Γιατί είναι κάπως παράδοξο να, να, να χρηματοδοτούμε το αποθεματικό της κρίσης για τους γεωργούς με τα κονδύλια της ίδιας της Γεωργίας. Αυτή πάντως ήταν η πρόταση για τη χρηματοδότηση του αποθεματικού κρίσης για τη Γεωργία. Τώρα για τα πιλωτικά προγράμματα, τα πειραματικά προγράμματα και σχέδια. Θα πρέπει να υποβληθούν, να γίνει μια αξιολόγησή τους από την Επιτροπή. Δεν θα αποφαθώ ε, επί των σχολείων και των σχεδίων. Άκουσα πολλές ε, καλές προτάσεις που σχετίζονται και με την διαπαιδαγώγηση. Εγώ είμαι υπέρμαχος της ανάπτυξης της υπαίθρου. Πιστεύω ότι η αγροτική ανάπτυξη συμβάλλει στη συνοχή και είναι έκφανση της εσωτερικής αλληλεγγύης. Η γεωργία επίσης δημιουργεί θέσεις απασχόλησης. Θα πρέπει όμως να δει και τα άλλα προγράμματα των άλλων δημοσιονομικών γραμμών. Γιατί όχι και ορίζοντας 2.000, έρευνα. Και το κοινό στρατηγικό πλαίσιο εφαρμογή των ταμείων. Γιατί να μην αναζητήσουμε περισσότερη συμπληρωματικότητα του Γεωργικού Ταμείου με τα υπόλοιπα ταμεία. Και εγώ πάντως περιμένω και άλλα βάσιμα επιχειρήματα. Ήδη άκουσα πολλά καλά επιχειρήματα και σημείωσα τις φιλοδοξίες σας, τις οποίες και εστερνίζομαι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Δενανό. Ευχαριστώ. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο για την έκθεση αυτή. Διαπιστώνω ότι υπάρχει μεγάλη βούληση από το Συνολό των Συναδέλφων να καταπολεμήσουμε τη γραφειοκρατία και να εργαστούμε υπέρ της απλούστευσης. Νομίζω ότι στο θέμα αυτό συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό. Το δεύτερο σημείο έχουμε το λεγόμενο αποθεματικό κρίσης που αναφέρθηκε επανειλημμένος και ε, το που θα χορηγηθεί. Εγώ νομίζω ότι τα χρήματα προς ε, τους Γιουργούς θα έπρεπε να επανέλθουν στους Γιουργούς, όμως ε, θα πρέπει φυσικά να χρησιμοποιήσουμε κάθε περιθώριο. Θέλω να πω ακόμη ότι το θέμα της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας ε, δεν ε, αποκλείει τη στήριξη στις μικρές εκμεταλλεύσεις, ε, κυρίως σε ευαίσθητες περιοχές, όπως τις ορεινές περιοχές, τις άκρες απομακρυσμένες περιοχές. Θα πρέπει η γεωργία να μπορεί να είναι βιώσιμη και να μπορεί να διατηρήσει στη ζωή την αγροτιά. Αυτό θα πρέπει να διατηρήσουμε και να ενθαρρύνουμε. Εγώ λοιπόν συμφωνώ με όσους είπαν ότι πρέπει σήμερα να μην καταργούμε πλέον τις γεωργικές ενισχύσεις γιατί ε, αυτές στηρίζουν την αγροτική μας επικράτεια. Και Επίσης, για κάποια ίσονο σημασία θέματα, άκουσα το θέμα για τις τοπικές αγορές ε, και εγώ νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό, αλλά νομίζω ότι περισσότερο η τοπική αυτοδίκηση και τα κράτη έχουν ρόλο εκεί να συστήσουν αυτές τις αγορές ε, και επίσης όλοι δίνουμε μεγάλη προσοχή στο θέμα της αστάθειας ε, των τιμών. Φυσικά το θέμα του γάλακτος προκύπτει συνεχώς σήμερα, αλλά έχουμε τέτοια αστάθεια και σε πολλούς άλλους τομείς. Νομίζω ότι θα πρέπει σύντομα να βρούμε τρόπο να καταπολεμήσουμε την ασταθία αυτή. Δεν είναι απλό το ζήτημα, αλλά θα, θα μας επιτρέψει να έχουμε ασφάλεια ε, στον εφοδιασμό. Επίσης, άκουσα και τι είπε ο κύριος Νίκονσον, ο οποίος ε, είπε έλεος μην μειώνεται κι άλλο τον προϋπολογισμό για τη Γεωργία και θα συμφωνήσω. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, περαιτέρω διαδικασία. Μέχρι 7 Μαΐου προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. 7 Μαΐου, 12 το μεσημέρι. Ευχαριστώ τους συναδέλφους και τον καλεσμένο μας, τον κύριο Φερνάντες. Ευχαριστώ και το συντάκτη της γνωμοδότησης. Ολοκληρώσαμε το σημείο 6, 5 και 6 και περνάμε στο επόμενο. Σημείο 7 λοιπόν, η προάσπιση των χρηματοοικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ε, ο προσανατολισμός των ελέγχων της κοινή γεωργικής πολιτικής στις ε, επιδόσεις. Ο κύριος Γκίζεκε είναι ο συντάκτης γνωμοδότησης, αρμόδια καθήλη επιτροπή, επιτροπή ελέγχου προϋπολογισμού. Συντάκτης, ε, εισηγητής έκθεση είναι ο κύριος Σαρβάμα, τον γνωρίζουμε. Ε, η έκθεση είναι έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας με θέμα την πράσπιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Η Επιτροπή, η Επιτροπή Γεωργίας αποφάσισε να συντάξει γνωμοδότηση ε, με θέμα τη σχέση μεταξύ της γεωργικής δραστηριότητας και της ευθύνης στην εφαρμογή της κοινή γεωργικής πολιτικής. Τα τελευταία χρόνια η κοινή γεωργική πολιτική γίνεται πιο περίπλοκη και διαφοροποιημένη Έχουμε όλο και περισσότερες ε, και νέες ε, απαιτήσεις, ε, κατάργηση προηγούμενων κανόνων. Όλα αυτά δημιουργεί μεγάλη περιπλοκή, επιβάρηση του κόστους και δύσκολη καθιστά τη διενέργεια των ελέγχων. Στόχος είναι λοιπόν να προσανατολίσουμε τους ελέγχους περισσότερο στα αποτελέσματα και στις επιδόσεις αλλά καλύτερα θα μας τα πει ο εισηγητής μας, ο συντάκτης της γνωμοδότησης για την ακρίβεια, ο κύριος Γιάννης Γκίσεκε, στον οποίο και δίνω το λόγο, παρακαλώντας το να μας κάνει την παρουσίαση της γνωμοδότησής του. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ είμαι, εδώ, εδώ. Γεια σας. Η χθεσινή ακρόαση έδειξε ότι η περιπλοκότητα της κοινή γεωργικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ιδιαίτερως χωρίς όμως να έχει μειωθεί η γραφειοκρατία. Οι γεωργοί που πρέπει να δαπανούν πολύ περισσότερο χρόνο να υποβάλουν αιτήσει για τη διαχείριση των εκμεταλλεύσεών τους και αυτό αποτελεί τελικά τον κανόνα. Το κόστος για τους ελέγχους ε, βρίσκεται στα 4 δις ε, ευρώ των, σε επίπεδο κρατών μελών με μια τάση αυξητική, κυρίω για, λόγω της, ε, του greening. Το σύστημα έχει φτάσει στα ωριά του, είναι σαφές αυτό και υπάρχει ανάγκη να δράσουμε άμεσα. Οπότε χαίρομαι και το είπατε και εσείς Πρόεδρε ε, για την πρωτοβουλία αυτή του εισηγητού της, ε, της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού και του Επιτρόπου να απλουστεύσουν την ε, γεωργική πολιτική έτσι ώστε να μπορέσουμε να ε, δικαιολογήσουμε τα όσα κάνουμε σε επίπεδο πολιτική και για του φορολογούμενου και για του γεωργού. Το υπερβλοκότητα των συστημάτων ελέγχου έχει να κάνει με την υπερβλοκότητα των προποθέσεων. Για να απλουστευτεί το πρόγραμμα ελέγχων και να μειωθεί και η γραφειοκρατία για τα κράτη-μέλη, για τα θεσμικά όργανα και του γεωργού, θα πρέπει να απλουστεύσουμε τα δεδομένα τη κοινή γεωργική πολιτική. Οι γεωργοί βεβαίως ε, με αυτά τα περίπλοκα ζητήματα και τα γραφειοκρατικά ε, σημεία ε, υπερφορτώνονται και ουσιαστικά κάνουν λάθη που δεν θα έκαναν αν τα πράγματα ήταν πιο απλά. Και όλα αυτά βεβαίω μετά πρέπει να εξεταστούν και από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Οπότε έτσι μπορούμε να μειώσουμε το ποσοστό λάθο και να μειώσουμε και το κόστος που υπάρχει από αυτό η γεωργία από την ε, δική μου τη χώρα, από τη Γεωργία, την Κάτω Σαξονία, παραπονιούνται ότι υποβάλλονται σε πολλούς ελέγχους διαφορετικούς, οι οποίοι γίνονται σε διαφορετικά χρονικά σημεία. Και πραγματικά χάνεται η ροή. Ε, οπότε θα πρέπει να υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για το θέμα των ελέγχων, όπου όλες οι όλοι οι έλεγχοι θα γίνονται για την ίδια ε, εκμετάλλευση την ίδια χρονική στιγμή. Επίσης, μιλούμε για μια ετήσια εξέταση το Single Audit Scheme, έτσι ώστε οι γεωργοί να μην χρειάζεται και την ίδια χρονιά και από την Κομισιόν και να ελέγχονται και από την Κομισιόν και από το Ελεκτικό Συνέδριο. Πολλά λάθη λοιπόν θα μπορούσαμε να τα έχουμε αποφύγει και θα μπορούσαμε και στο μέλλον να τα αποφύγουμε, κυρίω ό,τι αφορά το e-government, ε, το θέμα δηλαδή του software, που μπορεί να μα βοηθήσει να ενισχύσουμε το δυναμικό που έχουμε. Θα ήθελα βεβαίω να σα θυμίσω και τη χθεσινή ακρόαση. Ο εμπειρογνώμονα από την Πολωνία μα είπε ότι αρχικά ε, υπήρχε ένα κόστος 100 ευρώ για μια αίτηση και μετά από το σύστημα εισαγωγής ε, το, ε, του IT ε, αυξήθηκαν τα κόστη αυτά κατά 38%. Αλλά τα τελικά τις νέες τεχνολογίες θα πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε για να μας βοηθούν, όχι για να μας δημιουργούν, να μας νέα προβλήματα. Δεν μπορούμε οι νέες τεχνολογίες να αφήσουμε να, να κάνουν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες ακόμη πιο γραφειοκρατικές. Αυτά λοιπόν για τη δική μου γνωμοδότηση. Βεβαίω είμαι ανοιχτό στα σχολιά σα και χαίρομαι και πολύ για τη συνεργασία που θα έχουμε με τον εισηγητή από την άλλη επιτροπή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δεκάστρο πρώτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ παρεμβαίνω εκ μέρους των αδελφών ε, Πορσάνη που είναι ασκιώδης ηγητής εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και δεν μπορεί να συμμετέχει σήμερα στη συζήτηση εδώ αλλά φυσικά είναι διαθέσιμος για οποιαδήποτε ανταλλαγή σχολείων ε, φυσικά και κατόπιν της σημερινής ανάλυσης της πρότασης. Ο κύριος Τζανί ήθελε να υπογραμμίσει κάποιες επιτυχίες που εγώ θα παρουσιάσω τώρα καταρχήν ε, αναφέρεται στο ότι η μείωση της γραφειοκρατίας είναι αναγκαιότητα που όμως δεν θα πρέπει να ανοίξει το δρόμο στην αύξηση της απάτης. Γι' αυτό χρειάζεται μια προσέγγιση ολοκληρωμένη προκειμένου να είναι το σύστημα όσο το δυνατόν πιο στεγανό. Υπάρχει ένας μηχανισμός ελέγχου της κοινή αγροτικής πολιτικής ε, που έχει αρμοδιότητες σε διάφορα επίπεδα και σε εθνικό επίπεδο κεντρικές αρχές, οργανισμούς πληρωμών, οργανισμοί πιστοποίησης κτλ. αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως ελεκτικό συνέδριο και κομισιόν αυτό το σύστημα δημιουργεί υπερβολικό άχθος ε, για τους Ευρωπαίους εργοτές και γι' αυτό θα μπορούσαμε να έχουμε ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρος με ε, την απλοποίηση του λογαριασμού. Το δικαιωτικό άχθος ε, θα πρέπει να είναι ευέλικτο προκειμένου να αποφύγουμε πολύ ψηλά ποσοστά σφάλματος που οφείλεται στην μη δυνατότητα να ικανοποιηθούν αυτές οι απαιτήσει πλήρως και σε ό,τι αφορά τις άμεσες ενισχύσεις, συνολικό μπλοκαρισμά τους και ακόμη και σε περίπτωση που μπορεί να ανακύπτουν κάποια κρίσιμα στοιχεία σε ό,τι αφορά ένα τμήμα ε, της επιφάνειας. Αυτό παραμένει αμφισβητήσιμο και το πέρασμα σε ένα σύστημα ελέγχου που θα βασίζεται περισσότερο στις επιδόσεις θα πρέπει να συνεχίσει να είναι ο κύριος στόχος. Παρ' όλα αυτά, ο εισηγητής μας θεωρεί ο σκιώδης εισηγητής θεωρεί ότι θα πρέπει να ε, επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένους στόχους που θα είναι και δυνατό να υλοποιηθούν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Χόισλινγκ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τις ιδέες του. Πρέπει όμως ε, να διαφωνήσω με κάτι το ότι οι γεωργοί ασχολούνται με θέματα ελέγχων και κάθονται σε γραφεία και συμπληρώνουν αιτήσει. Ε, τι να σα πω, δείξτε τους με εμένα αυτού τους γεωργού. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Οι περισσότεροι είναι στα, στα χωράφια τους και ασχολούνται με αυτό. Είναι νομίζω ένας μύθος που κυκλοφορεί αυτό. Ε, υπάρχει μια αιτήση για την στρωματική ενίσχυση. Αν δεν καταφέρει να την, κάνει, να την ολοκληρώσει σε μία μέρα, Εντάξει, τότε όντω έχει πάρα πολλή δουλειά. Αλλά τώρα τι να πω, ότι αυτό συμβαίνει γενικώ και για όλου, δεν νομίζω. Πρέπει λοιπόν να το δούμε. Πρέπει να είμαστε και αξιόπιστοι προ τα έξω. Ε, αν τώρα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο το μισό του των εσόδων ε, ε, έρχεται από τον τομέα αυτό, έχουμε την υποχρέωση να το εξετάσουμε και να δούμε πού πάνε τελικά τα χρήματα αυτά. Δεν μπορούμε να αντιδρούμε έτσι εν θερμό και να πούμε όλα είναι πάρα πολύ δαπανηρά και χρονοβόρα ε, και στο τέλο ε, τι θα γίνει, δηλαδή οι γεωργοί θα μα στείλουν τον αριθμό του λογαριασμού του και θα του στέλνουμε εμεί τα λεφτά κατευθείαν. Χρειαζόμαστε ένα καλό μέτρο, ένα καλό μέτρο ε, για τι ε, πληρωμές και ένα καλό τρόπο ελέγχων. Βεβαίω θα πρέπει οι έλεγχοι να γίνονται από κοινού, να ελοκληρωθούν, να ενσωματωθούν, αυτό συμφωνώ. Είναι σκόπιμο να γίνει και νομίζω σωστό που το προτείνετε. Πρέπει βεβαίω να δούμε Πώ μπορούν να συνεργαστούν και μεταξύ του οι αρχέ που θα κάνουν του ελέγχους. Ε, χτες στην εισήγηση το είπα για την απλούστευση, ε, δεν το είπατε εσεί τώρα, αλλά τα περιβαλλοντικά μέτρα δεν νομίζω ότι είναι ο βασικός ε, λόγος για την ε, ύπαρξη γραφειοκρατίας. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που προκαλούν γραφειοκρατία. Ε, δεν είναι μόνο η αιτία τα, τα περιβαλλοντικά μέτρα. Τώρα, για το ελεκτικό συνέδριο νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Ε, έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις και οι, συντονιστέ και ε, συντονιστές επίσης με το ελεκτικό συνέδριο, οπότε νομίζω ότι μπορούμε και εμείς να παρέμβουμε στα πλαίσια της αρμοδιότητας που έχουμε. Πολλά πράγματα που ε, παρουσιάζονται στο κοινό είναι όντως ε, ίσως ε, λεπτομέρειες που τελικά μετατρέπονται σε πολύ μεγάλους ε, μύθους για σκάνδαλα κλπ. Επίσης, δεν θα πρέπει να έχουμε τον πρώτο πυλώνα στον πυρήνα τη σκέψης μας, αλλά τα μέτρα του δεύτερου πυλώνα για την γραφειοκρατία. Μέτρα δηλαδή που ναι, μπορεί να είναι πολύπλοκα, αλλά θέλουμε να τα ε, απλουστεύσουμε. Για, για τον πρώτο πυλώνα δεν νομίζω ότι είναι αυτό τελικά το, το πρόβλημα. Νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στα μέτρα του δεύτερου πυλώνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επιτέλους ε, έχετε τη θέληση να απλουστεύσετε την ΚΑΠ και να μειώσετε τις ταλαιπωρίες των γεωργών που χάνουν και χρόνο και χρήμα. Και δείχνει με έλλειψη σεβασμού ε, η μέχρι τώρα κατάσταση προς τον Γεωργό ε, που βλέπει τον ε, ελεγκτή να καταφθάνει έφνης. Εγώ που είμαι Γεωργός έχω αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα και μάλιστα ήρθε ένας ελεκτής ε, την ώρα που είμαι στο χωράφι μου. Είναι ταπεινωτικό, εξευθυλιστικό κάτι τέτοιο. Ενώ διαβάζουμε ότι 4 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν κατασπαταληθεί λόγω του υπερβολικού διοικητικού άχθους. Αυτό πραγματικά είναι άνω ποταμών. Ευχαριστώ κύριε Μαγκίνες. Uh, Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Πολλά στοιχεία της έκθεσης μπορούμε να τα υποστηρίξουμε. Νομίζω το σημείο 3 είναι το πιο σημαντικό και το δεύτερο κομμάτι αυτής της παραγράφου εκεί που λέει ότι ε, θα πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις στην βασική νομοθετική πράξη. Όπως είπε και ο Επίτροπος δεν είναι σε θέση να το κάνει αυτό, αλλά ένας από τους, το, ε, από τους ε, τομείς όπου έχουμε τα περισσότερα παράπονα από τους γεωργούς είναι ακριβώς η αυστηρότητα των ποινών. Για παράδειγμα, αν ένας γεωργός υποβάλλει την αίτησή του και υπάρχει, γίνει μια, ένας έλεγχος που δει ότι πάνω από 20% της ε, επιφάνειας της ε, εκμετάλλευσης ήταν ε, μη επιλέξιμη, αυτό σημαίνει ότι μειώνεται η άμεση πληρωμή του. Οπότε πρέπει να, κάποια στιγμή να μπορούμε να παρέμβουμε και στην βασική πράξη αν θέλουμε όντω να λύσουμε το πρόβλημα των εισαυστηρότητας των ποινών που επιβάλλονται στους, παραγω... στους γεωργούς. Το σημείο 6 επίσης είναι ενδιαφέρον για τα διάφορα κράτη-μέλη αλλά νομίζω ότι όταν οι χώρες έχουν πρόβλημα χρειάζονται βοήθεια με την εφαρμογή της νομοθεσίας, έτσι ώστε οι γεωργοί τους να μπορούν να συμμορφωθούν. Και σε ό,τι αφορά τώρα το e-government, είναι σημαντικό ε, όταν υπάρχει broadband, όταν υπάρχουν ε, δίκτυα. Ε, αυτό δεν γίνεται παντού όμως και επίσης ε, για πολλούς γεωργούς είναι δύσκολο να χρησιμοποιήσουν το e-government και πρέπει να έχουν και πρόσβαση επίσης είτε σε κάποιες, ε, κάποια συστήματα συμβουλευτικής, ε, κρατικά ή τέλος πάντων κάποιου είδους ε, βοήθεια για να μπορέσουν να συμπληρώσουν την αίτησή τους αν δεν μπορούν να το κάνουν μόνοι τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Φλάναγκαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω. Φαίνεται ότι οποιοδήποτε θέμα συζητάμε ε, στις τελευταίες 24 ώρες ανακύπτει το θέμα της απλοποίησης και περισσότεροι θέλουν εδώ να δουν απλοποίηση, όμως ε, φαίνεται ότι υπάρχει και μία σύγχυση ε, και εγώ το θεωρώ ότι είναι παράξενο γιατί εφόσον είμαστε δημοκρατικά εκλεγμένοι θέλουμε κάτι να γίνει και πάλι από ό,τι φαίνεται είναι αδύνατον. Τώρα, σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ένα περιβάλλον όπου θα δίνονται κίνητρα στους γεωργούς ε, να ε, σέβονται ε, τους κανόνες, μειώνοντας τους ελέγχους και φυσικά θα πρέπει να δοθούν τέτοια κίνητρα και σε επίπεδο κρατών μελών και να έχουμε ξεκάθαρες κατευθυντήριες γραμμές για τις κυβερνήσεις για να μειώσουν την πολυπλοκότητα των καθεστώτων, κυρίως μέσω ε, του Ταμείου Αγροτική ανάπτυξη. Ε, και αναφέρθηκε και κάτι πολύ καλό, ε, δηλαδή για το ότι σε ορισμένε περιπτώσει, μέχρι και το 100% των ενισχύσεων είναι ε, ποσό που πρέπει να πληρωθεί σε πρόστιμο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να επιβάλλονται πρόστιμο, όμως θα πρέπει καταρχήν να ξέρουμε τι σημαίνει συμμόρφωση, ε, ποιος είναι ο ορισμός του συμμορφούμε και στο επίπεδο ε, κράτους μέλους. Εγώ προέρχομαι από την Ιρλανδία και μπορώ να σας πω ότι εκεί υπάρχει τεράστια σύγχυση, γιατί φυσικά όταν σου επιβάλλεται ένα πρόστιμο και δεν ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, είναι πραγματικά τραγικό, γιατί δεν καταλαβαίνεις ξέρεις για ποιο πράγμα σου επιβάλλεται πρόστιμο και είναι εντελώ άδικο. Ευχαριστώ κύριος Ντόρφμαν. Ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. οι κανόνες της κοινή γεωργικής πολιτικής έχουν γίνει πιο πολύπλοκοι, δεν έχει μειωθεί η γραφειοκρατία και βέβαια αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει στο μέλλον. Η έλεγχοι κοστίζουν. Πρέπει να δαπανίσουμε, μάλλον δαπανάμε περίπου 40 δισεκατομμύρια και με την εισαγωγή του greening έχουν αυξηθεί και οι έλεγχοι. Οι νέε απαιτήσει σημαίνουν ότι έχουμε και μεγαλύτερο άχθος για τους γεωργούς. Η νέα ΚΑΠ θα πρέπει να γίνει λιγότερο γραφειοκρατική και θα πρέπει να υπάρχει απλούστευση. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, να προσφύγουμε στα βήματα που έχουν αναφερθεί στην έκθεση. Αυτό το καλωσορίζουμε και θα πρέπει να έχουμε και πιο αξιόπιστα δεδομένα στα κράτη-μέλη για να μπορούν να επαναλαμβάνονται οι έλεγχοι. Θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι με έναν τρόπο που να συνάδει με το ποσοστό σφάλματος. Επίσης, πάρα πολλοί γεωργοί ε, σήμερα δυσκολεύονται πάρα πολύ γιατί είναι τόσο γραφειοκρατικό το σύστημα και χρειάζονται παροχή συμβουλών. Βέβαια, αν προβαίναμε σε πλούστευση, αυτό θα σήμαινε ότι ε, θα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα και τα χρήματα του φορολογούμενου. Θα πρέπει να κάνουμε τους ελέγχους ε, να βασίζονται στον ε, κίνδυνο, δηλαδή να έχουμε μια προσέγγιση που να συνάδει με τον κίνδυνο, θα πρέπει οι γεωργοί να μην εκτίθενται σε δυσανάλογους ελέγχους. Έχουμε δαπανίσει πάρα πολύ χρόνο για να παρέχουμε κατευθυντήριες γραμμές ε, στους γεωργούς και βρίσκουμε πολύ μικρά λάθη και τους ποινικοποιούμε. Θα πρέπει να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη στάση και προσέγγιση απέναντι στους ελέγχους. Θα πρέπει όλοι οι έλεγχοι σε μία εκμετάλλευση να γίνονται ταυτόχρονα και θα πρέπει να επιμερίζεται ισομερός το άχθος για τους γεωργούς. Αντί να παίρνουν ε, τα χρήματα οι σύμβουλοι, οι γεωργοί θα έπρεπε να έχουν περισσότερο χρόνο να κάνουν τη δουλειά τους. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας ε, στον τομέα της γεωργίας. Θα πρέπει να εστιάσουμε αλλού προκειμένου να μην δεπανούμε το χρόνο μας με τον τρόπο αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σκοτ. Ευχαριστώ. Εμείς οι πράσινοι δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να αφήσουμε τη Γεωργία έρμα στις δυνάμεις της ελεύθερης ε, αγοράς. Ε, γιατί θα επικρατήσουν έτσι οι πολυεθνικές και θα φημώσουν και θα οδηγήσουν στη χρακοπία της οικογενειακής εκμεταλλεύσεις. Επίσης θα πρέπει να εξυπηρετήσουμε την Ήπεθρο. Επενδύουμε στη Γεωργία και στην Ήπεθρο και περιμένουμε κοινωνικά και ε, περιβαλλοντικά ωφέλη. Και αν θέλουμε να κρατήσουμε την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε σωστό έλεγχο των δαπανών μας, ιδιαίτερα της κοινής γεωργικής πολιτικής που είναι 43% του κοινοτικού πληθυσμού. Ε, θα πρέπει να δούμε τι πραγματοποιούμε για τις γεωργικές κοινότητες. θα πρέπει να έχουμε αποτελεσματικούς ελέγχους χωρίς να θυσιάζουμε τους, κα, τους στόχους του κανονισμού. Επίσης, ε, χρειάζονται και κυρώσεις. Οι κυρώσεις όμως δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ε, το επιχείρημα για την αναθεώρηση των ελέγχων είναι το κόστος του το υπερβολικό. Αλλά αυτό το 100% του συνολικού κόστος για τους ελέγχους δεν είναι υπερβολικό. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια σαφήνεια για τους γεωργούς, γιατί είναι άδικο να κάνουμε ελέγχους όταν δεν ξέρουν οι γεωργοί τι ελέγχεται. Και θα πρέπει ε, να γίνονται οι αιτήσεις από τους γεωργούς και οι έλεγχοι από τους επιθεωρητές. Θα ξέρουν τι να περιμένουν οι γεωργοί. Επίσης, ε, μεγαλύτερη σαφήνεια για τον όρο «ενεργός γεωργός». Δεν θέλουμε να ε, χρηματοδοτούμε πλούσιους γεωκτήμονες ή πλούσιους που απλώς αγοράζουν ε, μεγάλα αγροτεμάχια και δεν ασχολούνται με τη γεωργία. Ε, θα πρέπει να στηρίξουμε τους γεωργούς που καλλιεργούν, όχι τους ε, γεωκτήμονες. Θέλουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των ελέγχων και υψηλέ προδιαγραφέ των ελέγχων και επιθεωρήσεων. Αυτό περιμένουν και οι Ευρωπαίοι πολίτε για να βεβαιωθούν ότι τα κονδύλια του πιάνουν τόπο και ότι στηρίζουν τη γεωργία, μια γεωργία που είναι ευαίσθητη στι κοινωνικέ και περιβαλλοντικέ προτεραιότητε. Επίση, θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη επικοινωνία με του γεωργού για το πρόγραμμα οικολογικού προσανατολισμού και τα περιβαλλοντικά ωφέλη. Όπως είπαμε, το Ελεκτικό Συνέδριο προτείνει τα μέτρα πολλαπλής ε, συμμόρφωσης να ε, μετατραπούν σε καταμετρήσιμους ε, σκοπούς. Συμφωνούμε με αυτό. Καταλαβαίνουμε τη ματέωση των γεωργών από τους επανειλημμένους ελέγχους, αλλά είμαστε υπέρ ενός μεστού και ρωμαλαίου συστήματος ελέγχου και θέλουμε νέο λογιστικό έλεγχο που θα εφαρμόζεται συνεπώς ε, και θα εξηγείται δεόντως στους γεωργούς ώστε να ξέρουν ποιο είναι το σύστημα πριν ε, υποστούν ε, τα πρόστιμα και τις ποινές επειδή το παραβίασαν. Σας ευχαριστώ. Κύριος Νταντάν. Ο κύριος Νταντάν. Ευχαριστώ. Δεν το κατάλαβα ότι μου δίνατε το λόγο. Θα πρέπει να κάνουμε διαχωρισμό δύο τεινών εδώ. Έχουμε φενός ε, την πραγματικότητα, τον ελέγχο, την αποτελεσματικότητα και τον τρόπο διεξαγωγής τους. Και θα πρέπει φυσικά να έχουμε πιο ανθρώπινους ελέγχους και πιο απλούς ελέγχους. Θα πρέπει να τους ομαδοποιήσουμε και να τους συγχωνεύσουμε. Γιατί όλοι έχουμε παραδείγματα ελεγκτών, ε, άσχετα από που προέρχονται, που συμπεριφέρονται σαν ράμπο και όχι σαν ελεγκτές ενός ε, επίσημου οργανισμού, κάτι τέτοιο είναι παράδεκτο. Επίσης υπάρχει και το θέμα της απλούστευσης. Στο θέμα της απλούστευσης ε, ε, σας ομολογώ ότι αισθάνομαι κάποια δυσφορία. Ας μην ξεχνούμε ότι εμείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε καταθέσει 8.000 τροπολογίες στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν εξετάσαμε τα τέσσερα κείμενα. Και αυτές οι 8.000 τροπολογίες των Ευρωβουλευτών δεν συνέλαβαν ιδιαίτερος στην απλούστευση του κειμένου που ισχύει σήμερα. Οπότε θα πρέπει να αναλάβουμε και εμείς τις ευθύνες μας, αντί να κατηγορούμε άλλους και να είμαστε και ρεαλιστές. Ένα άλλο προβληματικό θέμα είναι ότι σε σχέση με το κείμενο που ψηφίσαμε, έχουμε κάποιες διαφορές ε, στην εφαρμογή να γίνει μια διευκρίνηση, αποσαφήνιση. Ποιος φταίει. Τα κράτη, οι εθνικές αρχές, οι περιφερειακές αρχές, οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτός ο υπερθεματισμός μεταξύ των γενικών διευθύνσεων, εκείνων που δεν έχουν προπολογισμό αλλά επιβάλλουν κάποιες απαιτήσεις στη γεωργική πολιτική, γιατί μερικές φορές ε, δεν αναγνωρίζουμε το κείμενο που ψηφίσαμε και την εφαρμογή του στην πράξη. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας. Για το φθινόπωρο έχουμε προγραμματίσει πολλές, ημερήσεις, ε, πολλές ε, συγγνώμη, δημόσιες ακροάσεις για να αναλύσουμε όλα αυτά τα θέματα, να δούμε τι προσθέθηκε στο διάστημα που μεσολάβησε από την ψηφοφορία μέχρι την έμπρακτη εφαρμογή του νομοθετικού κειμένου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντως, συμφωνήσαμε με την, ε, ε, για την ε, μεταρρύθμιση, ήμασταν υπεύθυνοι από πλευράς Κοινοβουλίου, θέλουμε όντως να μειώσουμε την γραφειοκρατία, αλλά πρέπει να μας βάλουμε τελικά βαθμό κάτω από τη βάση. Δεν τα έχουμε καταφέρει, δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά η γνωμοδότηση είναι πολύ σημαντική, γι' αυτό ασχολούμαστε με αυτή και χαίρομαι που τη συζητούμε σήμερα, γιατί χρειαζόμαστε μείωση της γραφειοκρατίας, και είμαστε τώρα σε ένα φαυλοκύκλο. Ο συνάδελφος είχε, είπε και πριν ότι θέλουμε ε, λιγότερους ελέγχους ε, γιατί ε, πάνε κάποιοι στι στις εκμεταλλεύσεις και ελέγχουν και οι γεωργοί δεν ξέρουν τι ελέγχεται και πάντα βρισκόμαστε σε ένα φαυλοκύκλο. Πρέπει όμως να υπάρχουν έλεγχοι. Αν υπάρχουν περισσότερα λάθη, το σύστημα αυτό που κάνει είναι να απαντάει με περισσότερους ελέγχους. Γι' αυτό πρέπει να μειώσουμε τη γραφειοκρατία. Και αυτό σημαίνει να εξασφαλίσουμε ότι το σύστημα δεν θα μπορεί να τύχει ε, παραποίησης. Έτσι ώστε να μπορούμε τελικά όντως να μειώσουμε στο τέλος και τους ελέγχους. Το είπε και ο συνάδελφος Χόισλινγκ. Υπάρχουν και στο πρώτο, στον πρώτο πυλώνα προβλήματα. Βάλαμε το greening. Εγώ νομίζω ότι δεν ανήκει στον πρώτο πυλώνα, επιδίνωσε την κατάσταση σε ό,τι αφορά του ελέγχου στο greening. Ούτω ή άλλω τι ε, άμεσε πληρωμέ μόλι το Δεκέμβρη μπορούμε να τι ε, κάνουμε. Έχουμε το greening εν τω μεταξύ. Και οι γερμανικέ αρχέ λένε ότι θα πρέπει και το Φεβρουάριο όμω να ελέγξουμε αν ακόμα το greening υπάρχει. Και τι θα γίνει τελικά, τι θα ελέγξουμε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ε, να να δούμε τι γίνεται στον έλεγχο, α πούμε, στι 10 Φεβρουαρίου. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα ε, ξεκαθαρίσουμε. Παρ' όλα αυτά μπορούμε ε, να έχουμε αυτό το βασικό, τη βασική επιδότηση, η οποία ναι είναι μια μείωση της γραφειοκρατίας, ε, μια τιμή, ένα εκτάριο, αυτό θα μπορούσε ίσως να είναι ένα βήμα προς τη μείωση της γραφειοκρατίας. Τρίτη παρατήρηση θα πρέπει να είμαστε θαραλέοι στον τρόπο που προχωράμε. Ξέρω ότι ο Επίτροπο είπε ότι θέλει να μειώσει τη γραφειοκρατία και αυτό. Αλλά δεν μπορούμε να αγγίξουμε τη βασική πράξη εν τω μεταξύ. Συζητούμε όμω διάφορες προτάσεις. Εγώ θα ήθελα να υπάρχουν πολύ ευρείε προτάσεις. Δεν ξέρω, κάποια στιγμή θα γίνει ένα mid-term review, θα γίνει ένα health check, κάτι θα γίνει, αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε. Εύχομαι λοιπόν μεγάλη, ε, καλή επιτυχία στον ε, εισηγητή και στου ε, σκιώδει εισηγητέ και εγώ βεβαίω θα του υποστηρίξω. Ελπίζω να έχουμε όντω καλέ προτάσει. Κυρία Μαγκίνε και πάλι. Ευχαριστώ. Και συγγνώμη που ξαναζήτησα το λόγο. Ξέχασα πριν να αναφερθώ στο χάρτη δικαιωμάτων των γεωργών. Δεν ξέρω αν ισχύει τέτοιο χάρτη ε, δικαιωμάτων των γεωργών σε όλε τι χώρε μέλη. Πάντω στην Ιρλανδία έχουμε ένα τέτοιο χάρτη. Θέλει επικαιροποίηση όμω. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν ε, μιλήσαμε στο ΕΛΚ, ζήτησε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Δικαιωμάτων των Γεωργών. Για να γίνεται σεβαστή η αξιοπρέπειά του όταν συμμετέχουν σε διάφορα συστήματα. Και επίση να αποσαφηνηθεί ο ρόλο των επιθεωρητών, των ελεκτών, τα ένδικα μέσα, μηχανισμοί προσφυγής και πώς να αντιμετωπίσουν οι γεωργοί την ε, γραφειοκρατία. Θα μπορούσαμε λοιπόν ε, μέσω των τροπολογιών μας προς αυτή την κατεύθυνση να σμπρώξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Σίγουρα θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Ο κύριος Ντες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Άκουσα πολύ προσεκτικά όλες τις παρεμβάσεις και τις ε, περισσότερες μπορώ να συμφωνήσω. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Πρέπει να πω κάτι όμως. Δυστυχώς δεν ε, ήταν ε, δυνατό στην προηγούμενη θητεία να δούμε το θέμα του greening που μπήκε στον πρώτο πυλώνα. Αν το greening είχε μπει στο δεύτερο πυλώνα, με βεβαίω την πρικοδότηση που του χρειάζεται, ίσως θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μεγαλύτερη ε, μείωση της ε, γραφειοκρατίας. Δυστυχώς δεν έτυχε πλειοψηφία η πρόταση αυτή και δεν έγινε. Τώρα η Κομισιόν ε, θέλει όντως να καλύψει τα κενά που υπάρχουν, να οδηγήσει όντως σε μείωση της γραφειοκρατίας και μέσω των κατεξοδοτήσεων πράξεων βεβαίω τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο και νομίζω ότι υπάρχει ευθύνη όλων μας για αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα τους ελέγχους, ένα είναι σαφές και θα συμφωνήσω με αυτό που είπαν πολλοί συνάδελφοι για θα πρέπει όντω εκεί που δίνονται κρατικά χρήματα να γίνονται και έλεγχοι. Και έλεγχοι. Αλλά η έλεγχοι θα πρέπει να είναι πρακτική. αν ο γεωργός δεν καταλαβαίνει τι πρέπει να δείξει στον ελεγχτή ε, προφανώς ο έλεγχος δεν θα έχει κανένα νόημα. Μιλήσαμε και για το ελεγκτικό συνέδριο για το θέμα των ελέγχων μεταξύ ε, λάθων και απάτης. Εκεί όντως πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή. Αν όντως υπάρχει απάτη, ναι, πρέπει οι ποινές να είναι αυστηρές. Ε, δεν πρέπει όμως να θεωρούμε ότι όλοι οι ε, ε γεωργοί ενσυνείδητα κάνουν απάτη. Υπάρχουν λάθη που δεν θα πρέπει, που δεν ουσιαστικά δεν επηρεάζουν τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων, δεν θα πρέπει να θεωρούνται λοιπόν να αυξάνονται κατα... Ε, αυτόματα και τα ποσοστά λάθους που καταγράφονται. Ο γείτονά μου ε, ε, είχε ένα... Πήγε, πήρε με κάποιο τρόπο πέντε μέτρα παραπάνω χωράφι από, από το γείτονα. Δεν το έκανε όμως επίτηδες, ούτε το κατάλαβε και δεν το δήλωσε. Και όταν έγινε ο έλεγχος ήρθαν και του είπαν ναι, λες δηλώνεις λιγότερο από ό,τι έχεις και αυτό καταγράφεται ως λάθος. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ε, ε, ή ως απάτη. Πρέπει να υπάρχει σαφής διαφοροποίηση λοιπόν μεταξύ των περιπτώσεων που όντως είναι απάτη και που όντως θα πρέπει να τιμωρούνται αυστηρά και των λαθών που δεν έχουν τελικά επιπτώσεις στον ευρωπαϊκό κορβανά. Κυρία Σλάιερ. Ευχαριστώ. Θέλω να υποστηρίξω το όσο είπε η κυρία Μαγκίνες. Αν ε, μιλάμε για την ΚΑΠ, αυτό είναι το ένα, αλλά πολύ συχνά Έχουμε υποψία από την πλευρά των ελεκτών, δηλαδή αντιμετωπίζονται οι γεωργοί σαν να είναι εγκληματίες που εργάζονται στο γεωργικό περιβάλλον. Εγώ νομίζω ότι αυτό συμβαίνει σε πολλές χώρες. Θα έπρεπε να σκεφτούμε και πολλά άλλα μέτρα που υπάρχουν. Μιλήσαμε για το θέμα της ευημερία των ζώων. Θα πρέπει οι γεωργοί να πληρώνουν σημαντικά τέλη όταν έρχονται ελεκτές. Αν δούμε τους κανόνες ε, για τα οικοσυστήματα ε, και γι' αυτό θα πρέπει να πληρώνουν οι γεωργοί. Έτσι λοιπόν ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι δεν υπάρχει επαρκής απλούστευση. Δηλαδή, οι γεωργοί δεν μπορούν να πετύχουν όλα όσα θα ήθελαν και φυσικά η δουλειά μας εδώ είναι να τους βοηθήσουμε. Ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ζητήσω συγγνώμη γιατί έφτασα καθυστερημένα Ξέρετε, είχαμε προβλήματα με τις πτήσεις. Όμως, ε, ευχαριστώ ε, τον συνάδελφο που παρουσίασε πάρα πολλές πτυχές ε, των αποψιών μας. Ξέρω ότι και στη σημερινή συζήτηση, αλλά και χθες, αναφέρθηκε το έγγραφο αυτό. Και νομίζω ότι αυτή η συζήτηση τώρα είναι σε πρώιμο στάδιο. Αυτό σημαίνει ότι και η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα παρουσιάσει κάποιες τροπολογίες στις αρχές Ιουνίου. Και νομίζω ότι εμείς έχουμε δυνατότητα να συζητήσουμε αυτά τα θέματα περαιτέρω εις βάθος. Τώρα, τι θέλω να ζητήσω από την Επιτροπή αυτή. Ότι θα έπρεπε να δώσουμε περαιτέρω χρόνο, ένα περαιτέρω μήνα, γιατί αυτή η προθεσμία θα μας επέτρεπε να κάνουμε καλύτερη δουλειά. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στο πλαίσιο αυτό. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Χόισλινγκ για δεύτερη φορά. Σύντομα παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε, σύντομα. Εντάξει, ο καθένα έχει ιστορίε που να σα πει για του ελέγχου που δεν πήγανε πολύ καλά ή που ελεγκτή ε, έλεγξε λάθο ελεγχόμενο. Εν πάση περιπτώσει όμω. Ε, συμφωνώ. Με του ελέγχου πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ε, να δούμε τι σημαίνει ακριβώ λάθο και τι σημαίνει απάτη. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Γιατί έτσι θα μπορέσουμε να καθαρίσουμε λίγο και τα, και τα στατιστικά. Καμιά φορά το θέμα του διαχωρισμού των, και του, της οριοθέτησης των εκμεταλλεύσεων δεν είναι θέμα απάτης, μπορεί να είναι θέμα του συστήματος. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει διαφοροποίηση και αυτό πρέπει να είναι σαφές. Και πρέπει να θέσουμε το σύστημα του ελέγχου σε τέτοια ε, κατάσταση έτσι ώστε να μπορεί να συμβουλεύει για να αποφεύγονται τέτοιου είδους λάθη. Να, υπάρχει, να δίνεται δηλαδή κάποιο είδους συμβουλή, κάποιο είδους βοήθεια για τα λάθη, για τα λάθη που γίνονται, έτσι ώστε να ελέγχεται και πώς συμπληρώνονται ας πούμε οι αιτήσεις κτλ. Πολύ γεωργοί ε, ε αισθάνονται και λίγο μόνοι τους όταν, ε, ή αποθαρρυμένοι όταν δεν, όταν δεν έχουν καμία βοήθεια από πουθενά. Ο ελεγχόμενος πρέπει και ο ελεγκτής πρέπει να ξέρουν τι ακριβώς θα ελέγξει και θα ελεγχτεί αντιστοίχως. Γιατί βεβαίως μιλούμε για ε, κονδύλια που πρέπει να δεσμεύονται από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Ευχαριστώ. Έχουμε μείνει πίσω στο χρόνο. Ο κύριος Φλάναγκαν και αυτός για δεύτερη φορά. Παρακαλώ. Χρόνου. Ναι, πολύ σύντομα. Δεν νομίζω ότι Πολύ συχνά έχουμε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από την ΚΟΥΕ της Πρεσίνους τις τελευταίες 24 ώρες. Ε, ε, ακούσαμε την πρόταση της κυρίας Μαγκίνες ε, για τη χάρτα δικαιωματών των εργατών. Την ίδια πρόταση έκανα και εγώ χτες και έλαβα πολύ θετικό feedback. Έτσι λοιπόν ρωτήσαμε πώς μπορούμε να το προωθήσουμε αυτό. Γιατί και βλέπω εδώ ότι συμφωνούμε σε κάτι, στην απλούστευση. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να κάνουμε κάτι απτό έτσι ώστε να έχουμε μια χάρτα δικαιωμάτων ε, για τον Ευρωπαίο αγρότη. Πώς μπορούμε να το προωθήσουμε γιατί βλέπω ότι υπάρχει συμφωνία. Ευχαριστώ και τώρα. Η κυρία Κριστίν Μπόλσμαν, εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Πολύ μιλήσατε για την απλούστευση και ξέρω ότι σας απασχόλησε και χθε το απόγευμα το θέμα αυτό. Γι' αυτό δεν θα επισέλθω σε πολλές λεπτομέρειες. Θα ήθελα να πω απλώς αυτά που έλεγε και ο Επίτροπος και η Επιτροπή. Με την απλούστευση των μέτρων απλουστεύονται και οι έλεγχοι. Ο τρόπος διενέργειας των ελέγχων αντανακλά την περιπλοκότητα των μέτρων. Και μια και είμαι αρμόδια για τον έλεγχο στη Γενική Διευθύνση Γεωργίας, τον λογιστικό έλεγχο στα κράτη-μέλη, θα ήθελα να σας πω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είπε ότι φυσικά δεν πρόκειται να γίνει η απλοποίηση ε, στην πλάτη της ε, νομικής πειθαρχίας και της χρηστής δημοσιονομικής πειθαρχίας. Το θέμα είναι ότι θέλουμε καλύτερους ελέγχους και όχι περισσότερους ελέγχους. Αυτός είναι ο κοινό μας στόχος από ό,τι κατάλαβα. Μερικοί αναφερθήκατε στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ που δαπανώνται για τον έλεγχο, όπως είπατε. Θα ήθελα να σας υπογραμμίσω ότι τα 4 δισεκατομμύρια αφορούν τον έλεγχο ε, με διασταλτική έννοια, δηλαδή την διαχείριση και τον έλεγχο είναι και το κόστος δηλαδή της ε, λήψης και επεξεργασίας των αιτήσεων ε, των γεωργών ώστε να μπορούν να πάρουν τα κονδύλια. Επίσης το κόστος των παροχής συμβουλών που παρέχουν οι φορείς πληρωμών. Ε, είναι ένα σύστημα που εξυπηρετεί και διευκολύνει τους αγρότες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους σωστά. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στο κόστος των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν λέω ότι το, το ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου και διαχείρισης και με το νέο σύστημα άμεσων ενισχύσεων δεν θα έχουμε περισσότερους ελέγχους. Πάντως εξετάζουμε εξονυχιστικά το κόστος κάθε μονομένης δράσης. Και η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και πάλι φέτος θα αποτιμήσει μαζί με τα κράτη-μέλη το κόστος της διαχείρισης και του ελέγχου, ώστε θα σας έρθει ένα ενημερωμένο ποσό μπορεί να είναι 4 δισεκατομμύρια, μπορεί και όχι. Και επίσης θα ληφθεί υπόψη η, με, εφαρμογή της μεταρρύθμισης και φέτος. Δεν έχουμε συγκεντρώσει ακόμη όλες τις πληροφορίες από τα κράτη-μέλη. Είναι μια διαδικασία που θα κρατήσει μέχρι το τέλος του έτους. Κάποια σχόλια για το σχέδιο γνωμοδότησης. Μερικοί αναφερθήκατε στην ανάγκη μείωση του αριθμού των ελέγχων επιτόπου στι γεωργικέ εκμεταλλεύσει. Αυτό ήδη γίνεται για τα κράτη-μέλη. Υπάρχει δυνατότητα των κρατών μελών να μειώσουν από 5 σε 3% του ελέγχου. Και αν ισχύει ένα ποσοστό σφάλματο κάτω από 2% και μάλιστα για δύο συναπτά χρόνια. Κάποιε χώρε ήδη όταν σημείωσαν ε, ποσοστά σφάλματος κάτω του 2% για δύο χρόνια μπόρεσε να μειώσει του ελεγχου από 5% σε 3% και μάλιστα από φέτος. Δεν υπάρχει σχετικό κανονισμός, είναι μια μεταβατική ρύθμιση. Οπότε υπάρχει αυτή η δυνατότητα μείωση των ελέγχων. Αλλά προϋποθέτει ε, ένα ποσοστό σφάλματο σφάλματος ε, κάτω του 2%. Γιατί είναι σημαντικό να ε, λειτουργούν αυτά τα συστήματα με χαμηλά ποσοστά σφάλματο. Μερικοί είπατε ότι ε, δεν θα πρέπει να ελέγχουμε τους γεωργούς που συμμορφώνονται. Μα γι' αυτό όλοι οι κανονισμοί ζητούν ανάλυση του κινδύνου. Και αν γίνει μια τέτοια ανάλυση του κινδύνου, ο έλεγχος δεν γίνεται που, των γεωργών που συμμορφώνονται, αλλά αυτών που υπάρχει κίνδυνος να μην συμμορφωθούν. Δεν γίνεται τυχαία επιλογή των γεωργών, αλλά επιλογή με βάση την ανάλυση κινδύνου. Επίση, συμφωνώ μαζί σα ότι θα πρέπει να δοθούν σωστέ κατευθυντήριε γραμμέ στου γεωργού, ιδιαίτερα με τη μεταρρύθμιση. Και έχουμε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη για να ισχύσουν τέτοιε κατευθυντήριε γραμμέ και προσανατολισμοί. Επίση, να αποσαφηνήσω ότι υπάρχει δυνατότητα μείωση των ελέγχων στο 3% αν το ποσοστό σφάλματο σε μια δεδομένη χώρα είναι χαμηλό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Δεκάστρο τώρα. Δεν θέλετε το λόγο. Ωραία. Οπότε ο εισηγητή μα, ο κύριο Γκίζεκε. Ευχαριστώ πολύ για τι πολύ επικοδομητικέ ε, παρεμβάσει σα. Ε, Χαίρομαι ότι υπάρχει από όλε τι ομάδε ε, συνένεση. Το θετικό είναι ότι μπορούμε με μια τέτοια γνωμοδότηση ε, να ε, ξεκινήσουμε και μια χάρτα για τα δικαιώματα των γεωργών, όπω είπε και η συνάδελφο. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό, αλλά δεν θέλουμε, να, θέλουμε να βελτιωθούν τα πράγματα για του γεωργού. Δεν θέλουμε να του θεωρούμε όλου απαταιώνε. Θέλουμε όμω όταν υπάρχει περίπτωση απάτη, να μπορούν να επιβληθούν ποινέ. Εγώ ευχαριστώ όλους ε, και τους σοσιαλιστές ε, που μου κάνανε πολύ συγκεκριμένε ε, προτάσεις. Αν μου τις στείλετε θα τις δεχτώ. Ευχαρίστω, είμαι ανοιχτό σε προτάσεις. Κύριε Χόισλινγκ, για το πόση γραφειοκρατία γίνεται, μένει τελικά στον, στον Γιώργο. Όντως, το greening έφερε από τον πρώτο πυλώνα πολύ μεγαλύτερη γραφειοκρατία. Χτε ε, οι εμπειρογνώμονε ε, μα είπαν ότι ασχολήθηκαν κάποιοι από αυτού με 20 χρόνια ε, με την Γεωργία και σήμερα οι Γεωργοί φοβούνται γιατί δεν ξέρουν τι πρέπει να εφαρμόσουν και τι όχι. Οπότε εμεί πρέπει να πλουστεύσουμε ως νομοθέτες τα πράγματα. Ο γεωργό πρέπει να ξέρει τι, πράγμα, τι πρέπει να εφαρμόσει και τι όχι. Χαίρομαι λοιπόν για τι τροπολογίε σα. Οι σοσιαλιστέ είπατε ότι θέλετε να αναβάλουμε για ένα μήνα την υποβολή των τροπολογιών. Θα είναι δύσκολο γιατί πρέπει να δώσουμε την γνωμοδότηση η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού και εκεί υπάρχουν συγκεκριμένε προθεσμίε. Οπότε πρέπει να το, να το στείλουμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τι ε, προθεσμίε. Οπότε είμαι λίγο διστακτικό να σα δώσω ένα μήνα παραπάνω. Ε, για με βάση και τα όσα είπατε, εντάξει, δεν θα έχουμε 8.000 τροπολογίε, υποθέτω. Ε, Ξεκινάμε με καλά παραδείγματα, έχουμε μια προθεσμία σύντομη. Α κάνουμε λοιπόν καλέ ε, τροπολογίε έτσι ώστε να καταλήξουμε και σε καλέ συμβαστικέ προτάσει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ γιατί είχαμε πολύ εμβριθεί και εμπεριστατωμένη συζήτηση που είμαι σίγουρος ότι θα εμπλουτίσει και τη δική σας γνωμοδότηση κύριε Γκίζικε. Όπω είπατε, η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών λήγει στι 7 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Αφιερώσαμε πολύ χρόνο στο πρόβλημα αυτό, αλλά είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Σημειώστε λοιπόν τις προθεσμίες και να περάσουμε στο επόμενο σημείο, το σημείο 8, που προβλέπει ανταλλαγή απόψεων με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα την παράταση της περίοδου επιλεξιμότητας των δαπανών για τα προγράμματα ανάπτυξη πέθρου για την περίοδο 2007-2013. Το Μάρτιο, μεγάλος αριθμός χωρών τάχθηκε υπέρ της πιθανότητας παράτασης της περίοδου Επιλεξιμότητα των δαπανών για προγράμματα ανάπτυξη υπαίθρου για την περίοδο 2007-2013. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε έτοιμη να εξετάσει το αίτημα αυτό που θα έπρεπε να επισημοποιήσει με μια νομοθετική πρόταση. Θέλουμε τώρα περισσότερη ενημέρωση για το θέμα αυτό. Ποια ήταν τα αποτελέσματα των εσωτερικών συζητήσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ποιες είναι οι προθέσεις της. Γι' αυτό και δίνω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για να μας ενημερώσει. Το λόγο του κύριος Μιχάηλ Ντουμίτρου, Διευθυντής στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Έχετε το λόγο, περιμένουμε πληροφορίες. Ε, Ευχαριστώ. Η Κομισιόν γνωρίζει ότι σε πολλά κράτη-μέλη οικονομικές ε, δυσκολίες ε, έχουν οδηγήσει σε πιο αργή εφαρμογή των προγράμματων γεωργικής ανάπτυξης στην περίοδο 2007-2013. Η Κομισιόν ε, κατανοεί τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτά τα κράτη-μέλη και εξετάζει την πιθανότητα να επιτρέψει την ολοκλήρωση των εφιστάμενων συμβάσεων και των πληρωμών κανονισμός επιτρέπει υπό συγκεκριμένε προποθέσει τη δυνατότητα να καλυφθούν όλες οι δαπάνε, δηλαδή δαπάνε αυτής της περίοδου από τι συνεισφορέ τη νέα περίοδου στο πρόγραμμα 2014-2020, δηλαδή για τι κρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων, αν επιλέξουν αυτή την οδό τα κράτη-μέλη, είναι δυνατόν να θα χρησιμοποιήσουν σε αυτή την περίοδο. Όπω ε, είπαμε, 11 κράτη-μέλη που υποστηρίζονται από άλλα 6 κράτη-μέλη έχουν ανανεώσει το αίτημα στην Κομισιόν για να προτείνουμε και να εισαγάγουμε έναν οργανισμό που θα έχουμε παράταση για 6 μήνες μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016 για την περίοδο επιλεξιμότητας ε, των απανών ε, στα πρόγραμμα για την περίοδο 2007-2013. Αυτά τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι η παράταση θα μπορούσε να είναι ο καλύτερος τρόπος για να χρησιμοποιήσουν στο δυνατόν καλύτερα τα κονδύλια που έχουν ήδη δεσμευτεί ενθαρρύνουμε τη χρήση όλων των υφιστάμενων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και φυσικά προκειμένου η Κομισιό να συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη για να βελτιστοποιηθεί η χρήση των πιστώσεων, ε, το Συμβούλιο θεώρησε ότι αυτό πρέπει να γίνει εντός της ευελιξίας ε, των σημερινών κανόνων. Αυτό ήταν ισχυρό πολιτικό μήνυμα. Η Κομισιόν κατάλαβε ότι θα πρέπει να σεβαστούμε, να μείνουμε εντός των κανόνων αυτών. Ε, ο νομοθέτης ε, τώρα δεν έχει δώσει εξουσία στην Κομισιόν να εισαγάγει την παράταση της περίοδου επιλοξιμότητας ε, για τα προγράμματα 2007-2013 η Κομισιόν έχει αναλύσει τις νομικές διατάξεις πολύ προσωπικά και κατέληξε ότι ο μόνος ε, νομικά εύρωστος τρόπος ε, θα απαιτούσε κανονισμό του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου που θα ακολουθούσε, θα την τακτική νομική διαδικασία. Όπως γνωρίζετε, η τακτική διαδικασία θα ήταν δύσκολο να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του έτους ακόμη και αν υπήρχε ισχυρή πολιτική δέσμευση από όλα τα θεσμικά όργανα. Η παράταση της περίοδου επιλεξιμότητας θα ήθελε επιπλέον δημοσιονομικούς πόρους που δεν έχουν προβλεφθεί από το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Το ε, Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ε, ε, είναι ένα από τα κυρία ταμεία. Θα πρέπει να δούμε και τις συνέπειες για τα άλλα δύο ταμεία μέχρι τώρα έχει αρνηθεί η Κομισιόν να προσφέρει την παράταση. Επίσης, η παράταση της περίοδου μέχρι το 2016 θα μπορούσε να αυξήσει την πρόσληψη του κονδυλίου και θα ήθελα να πω ότι στο εγγύς μέλλον ε, θα υπήρχαν πολύ λίγα προβλήματα για τα κράτη-μέλη, ενώ η προχρηματοδότηση για ένα, πρόβλημα, για ένα πρόγραμμα φτάνει το 95% η αποζημίωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σταματά και τα κράτη-μέλη μπορούν να συνεχίσουν ε, τις δαπάνες, αλλά θα πρέπει να χρηματοδοτούν τα πάντα από μόνο τους μέχρι να δοθούν τα υπόλοιπα χρήματα στο τέλος του προγράμματος. Στα τέλη του 2015 τα περισσότερα προγράμματα θα φτάσουν στο 95%. Έτσι λοιπόν η παράταση των 6 μηνών θα μετακινήσει τις τελικές πληρωμές 6 μήνες αργότερα και θα αυξήσει την ανάγκη για εθνικά κονδύλια κατά τη διάρκεια της περίοδου αυτής. Συνεπώς ο καλύτερος τρόπος να διασφαλίσουμε τη συνεχή ροή κονδυλίων στα κράτη είναι να εργαστούμε προς την υιοθέτηση και εφαρμογή ε, των νέων προγραμμάτων 2014-2020, όπου έχουμε ήδη τα νέα κονδύλια. Σήμερα, μετά από έκκληση από τα κράτη-μέλη, Κομισιόν αξιολογεί όλες τις πτυχές και την ε, δυνατότητα ε, υλοποίησης, ενώ είναι και σε στενή επαφή με τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη. Δεδομένης της φύσης της νομικής διαδικασίας, ε, ισχυρή υποστήριξη από τα κράτη-μέλη και θεωρούμε αυτό πρέπει να πάει πέρα από το Υπουργείο Γεωργίας, πρέπει να ε, μας παρασχεθεί για να πετύχουμε την υιοθέτηση μια τέτοια πρωτοβουλία μέχρι τα τέλη του 2015. Η Κομισιόν εργάζεται εντατικά για να ξεκαθαρίσει εσωτερικά ζητήματα που θα πρέπει να επιληθούν για το να αποφασίσει αν χρειάζεται να υλοποιηθεί μια τέτοια πρωτοβουλία. Η Κομισιόν συνεχίζει να συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη για οποιαδήποτε δυνατότητα ε, να βελτιστοποιήσει και να μεγιστοποιήσει τη χρήση των κονδυλίων ε, από την περίοδο 2007-2013. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ και ευχαριστούμε ιδιαίτερος γιατί ήταν πολύ σαφής και σύντομος. Ο κύριος Μπραν, ένα λεπτό παρακαλώ. Μία ερώτηση. Μία διευκρίνηση θα ήθελα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλοι γνωρίζουμε την απάντηση. Είναι μάλλον ρητορική ερώτηση. Μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε ότι κάτι τέτοιο δεν θα δημιουργήσει ε, ανάγκη για συμπληρωματικές δαπάνε. Δηλαδή αυτή η πρόταση δεν θα επιφέρει επιπρόσθετες ε, δαπάνες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λάμπεργκα. Ευχαριστώ. Ήμουν έτοιμος να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρωτοβουλία που ανέλαβε, ε, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία για πολλούς γεωργούς που αποφελούνται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δίνει την τέτοια σημασία στο ζήτημα αυτό. σαν να το κρίνει υποδιέστερο ή να θεωρεί ότι οι Υπουργοί Γεωργίες δεν ενδιαφέρονται. Μα 17 χώρες μέλη έδειξαν ενδιαφέρον. Δεν το γνωρίζουν αυτό οι Υπουργοί Γεωργίες. Πώς είναι δυνατόν να πιστεύετε ότι θα διαφωνήσουν. Επίσης, η αλληλεγγύη είναι μία από τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλοι γνωρίζουμε ότι στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε τους γεωργούς θα πρέπει α, να το κάνουμε όταν έχουν ανάγκη ιδιαίτερως. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι δικαιούχοι πολύ δύσκολα βρίσκουν συγχρηματοδότηση για διάφορα προγράμματα και σχέδια εξαιτία των τραπεζών σε μεγάλο βαθμό και της απροθυμίας τους για δανεισμό. Δεν φταίνει η γεωργοί. Οι τράπεζες φταίνε. Οπότε, οι τράπεζες για να είναι ασφαλείς ουσιαστικά παρεμποδίζουν τη διεξαγωγή κοινοτικών προγραμμάτων όταν απαιτείται στη χρηματοδότηση. Έτσι, οι γεωργοί θα χάσουν τα χρήματα που έχουν ήδη επενδύσει. Και εμεί αντί να τους στηρίζουμε και να προσπαθούμε να τους διευκολύνουμε, τους βάζουμε και κόμματα Το θέμα είναι να μπορέσουν οι Γεωργοί να συνεχίσουν τα προγράμματά τους και όχι ήδη να χάσουν αυτά που επένδυσαν. Φυσικά και θα πρέπει να επεκτείνουμε για άλλο ένα εξάμεινο την προθεσμία ε, ή την περίοδο επιλεξιμότητας των δαπανών. Επίσης, θα πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα των ανισορροπιών μεταξύ των διαφόρων γεωρικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα άλλο επιχείρημα υπέρ της παράτασης περίοδου επιλεξιμότητας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Νταντσίλα. Σας ευχαριστώ. Πιστεύω ότι θα πρέπει αυτό το αίτημα να μεταφραστεί σε νομοθετική πρόταση. Το είπε και από μόνη της Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι οικονομικές δυσχέρειες και αδειξότητες οδήγησαν στη μείωση των προγραμμάτων ανάπτυξης της υπαίθρου. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμόσουμε την πρόταση αυτή. Γιατί χάρη στην παράταση αποσοβείται ο κίνδυνος ε, να μείνουν εκκρεμή κάποια προγράμματα που ήδη έχουν ξεκινήσει στην Ήπεθρο και θα μπορέσουν και τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν προβλήματα να συνεχίσουν αυτά τα προγράμματα για μεγαλύτερη περίοδο. Στη συζήτηση του προϋπολογισμού για το 2016 μίλησαμε για την ανάγκη εδαφικής συνοχής και την ανάγκη ανανέωση των γενεών και ενθάρρυνση των νέων γεωργών να ασχοληθούν με τη γεωργία. Έχουμε την ευκαιρία με αυτή την νομοθετική πρόταση να περάσουμε από τα λόγια στα έργα και να υλοποιήσουμε την συνοχή. Την εδαφική συνοχή μεταξύ μετροπόλων και Υπέθρου, αλλά και την ε, συνοχή μεταξύ των γενεών. Επαναλαμβάνω αυτό το αίτημα το υπέβαλαν από κοινού 17 χώρες μέλη. Δώστε μια ευκαιρία στα σχέδια να συνεχιστούν, στα προγράμματα αυτά να συνεχιστούν και να μην κολλήσουν ιδιαίτερα σε ευαίσθητες περιοχές όπως είναι οι υπαίθριες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γουτσεφ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις πληροφορίες που μας υπέβαλε. Η περίοδος αυτή ε, και το αίτημα για την παράταση της, της περίοδου επιλεξιμότητας ε, ήταν ε, αίτημα που βρήκε πολύ γόνιμο έδαφος στο Συμβούλιο. Δεν υπήρχε ούτε μία αρνητική ψήφος και πολλές χώρες το ζήτησαν έντονα ακριβώς για να μην μείνουν στη μέση μερικά προγράμματα. Η παράταση της περίοδου επιλεξιμότητας θα επιτρέψει στους γεωργούς να ολοκληρώσουν σημαντικά προγράμματα στην Ήπεθρο. Ας μην ξεχνούμε ότι τα κονδύλια της ΚΑΠ είναι για πολλούς γεωργούς η μόνη πηγή εισοδήματος και η μόνη δυνατότητα να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Είναι κρίμα για διοικητικούς λόγους να μείνουν ατελείωτα ορισμένα προγράμματα. Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με δημιουργικό τρόπο και με αναθεώρηση του σχετικού κανονισμού να ε, δεχτεί το αίτημα και να παρατείνει την περίοδο επιλεξιμότητας. Η παράταση της περίοδου επιλεξιμότητας των δαπανών, κατά τη γνώμη μου, ε, δεν θα απαιτήσει συμπληρωματικά κονδύλια. Είναι απλώς μια χρονική παράταση. Ερωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρείτε ότι χρειάζονται επιπρόσθετα κονδύλια για την παράταση αυτή. Τέλος, θα ήθελα να σας θέρμα παρακαλέσω να μην τιμωρήσουμε τους γεωργούς που καλή την πίστη ήθελαν να ολοκληρώσουν τα προγράμματα αυτά. Θα πρέπει να πράξουμε τα δέοντα ώστε να υλοποιήσουμε τους στόχους της ΚΑΠ και να έχουμε μια πιο ανταγωνιστική γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Μπούντα. Uh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις uh, παρατηρήσεις σας. Καταρχάς, να ζητήσω από την Κομισιόν να μελετήσει και άλλα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν σε άλλους τομείς, όπου έχει υπάρξει όντως παράταση της ε, περίοδου επιλεξιμότητας. Γιατί εδώ δεν μιλούμε για έξτρα χρήματα, για έξτρα κονδύλια. Μιλάμε για χρήματα τα οποία έχουν δοθεί για συγκεκριμένους σκοπούς, αλλά δεν δαπανήθηκαν λόγω ε, γραφειοκρατίας. 17 κρατημέλη ζητούν αυτή την παράταση. Η Κομισιόν τι ακριβώς περιμένει. Γιατί δεν κάνει αυτό που ζητούν τα κρατημέλη. Και είναι 17, δεν είναι ένα και δύο. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο και πάλι στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απαντήσει, θα ήθελα και εγώ να επισημάνω ότι η οικονομική κατάσταση, η κρίση, οδήγησε στην ε, καθυστέρηση κάποιων προγραμμάτων. Και γι' αυτό δεν θα πρέπει με διαδικαστικό και διοικητικό τρόπο να στερήσουμε τη δυνατότητα αξιοποίηση αυτών των κονδυλίων. Θα πρέπει να επιτρέψουμε την σωστή διεκπαιρέωση των προγραμμάτων ανάπτυξη πέθρου. Είναι πολύ σημαντική και ε, ευάρεστη νομίζω αυτή η πρόθεση. Και μάλιστα δεν νομίζω ότι υπάρχουν και συμπληρωματικές δαπάνες λόγω της παράτασης της περίοδου αυτής. Τώρα θα δώσω το λόγο στον Διευθυντή της Επιτροπής Γεωργίας, της ε, Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, για να απαντήσει στις ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σημείωσα όλες τις ε, παρεμβάσεις, σημείωσα τις ενσυχίες των βουλευτών και βεβαίως θα τις ε, μεταφέρω στην Κομισιόν, στον Επίτροπο. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματα που μου τέθηκαν. Καταρχάς, για, το, extra, για τις έξτρα δαπάνες. Αν ε, ε παρατείνουμε την ε, περίοδο επιλεξιμότητας μπορεί να υπάρξουν νέα, νέες δαπάνες αλλά πάντα μέσα στα πλαίσια των ε, δεσμεύσεων που έχουμε για την περίοδο, περίοδο 2017-2013. Παρ' όλα αυτά η παράταση αυτή τη περίοδου τη επλεξιμότητα θα σήμαινε ότι αυτή η δαπάνη θα επιστροφεί από την Κομισιόν στα πλαίσια του νέου πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου. Οπότε θα χρειαστούμε έξτρα πόρους το 2017 για να ε, επιστρέψουμε αυτά τα χρήματα. Αυτή είναι η δημοσιονομική επιπλοκή ως προς αυτό. Τώρα, για τη συνέχιση των α, τρεχουσών συμβάσεων, όπως είπα και στην παρέμβασή μου, υπάρχουν δυνατότητες αυτέ ε, αυτές οι συμβάσεις να συνεχιστούν. Αλλά αυτή η δυνατότητα είναι είτε εντός των ορίων ή της παρατεταμένης περίοδου, αν το αποφασίσουμε, ή αυτή η δαπάνη μπορεί να καλυφθεί από τη συμβολή του EFRD ε, στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περίοδου εάν τα κρατη αποφασίσουν να πληρώσουν τις προϋποθέσεις για, την, ε, για αυτές τις νέες συμβάσεις στα πλαίσια των ε, νέων οικονομικών πλαισίων που θα υπάρξουν. Παίρνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας το γεγονός ότι 17 κρατη ζητούν να υπάρξει, ή μάλλον ανανεώνουν το αίτημά τους να υπάρξει επιλεξιμότητα και αυτό είπα ότι πρέπει να γίνει μέσω τη συνήθω διαδικασία, μέσω μια βασική πράξη και τώρα αξιολογούμε όλες τις δυνατότητες ε, σκοπιμότητας ε, για το κατά πόσο μπορεί να περάσει μια βασική πράξη και αν μπορούμε να, κάνουμε, να έχουμε μια τέτοια ε, πρωτοβουλία και να την ολοκληρώσουμε εντό του χρόνου γιατί αλλιώ δεν θα είμαστε εντό των χρονικών ορίων και θα είναι άσκοπο να γίνει όλο αυτό. Πρέπει να τα σκεφτούμε λοιπόν όλα αυτά, συμπεριλαμβανομένου και του γεγονότο ότι 17 κράτη-μέλη σημαίνουν πλειοψηφία των κρατών μελών αλλά όχι απόλυτη πλειοψηφία σε όρους πληθυσμιακούς. Οπότε ε, δεν έχουμε ακόμη τα όρια που υπάρχουν, που τίθενται ως προς αυτό. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε για τις απαντήσεις και τα σχόλιά σας. Νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπέρ της παράτασης της περίοδου επιλεξιμότητας. Οπότε συμφωνούμε. Θα περάσουμε σε λίγο στις συνεδρίες των συντονιστών. Ε, στις 3 θα ψηφίσουμε, γι' αυτό μην ξεχάσετε τις ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας. Ολοκληρώνεται η τακτική ε, συνεδρία Επιτροπής η πρωινή, μια σύντομη διακοπή και θα επανέλθουμε στις συνεδρίες των συντονιστών.